Παρακαλώ στις θέσεις σα όλοι. Θα ήθελα να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία τους όλους τους Γερμινείς και τις Γερμινείς. Πριν τώρα να ξεκινήσουμε αυτή την ομάδα εργασίας ε, για το πώς επηρεάζουν τα πράγματα, τα γεωργικά και τα αγροδιατροφικά, θα ήθελα να σας ενημερώσω σύντομα πάνω στο ε, ε, θέμα ποζέι της Τετάρτης να σας πω ότι αυτό το θέμα θα είναι στην ημερήσια διάταξη για τη σύνοδο την επόμενη εβδομάδα και ο κύριος Άλβες, ο εισηγητής, δεν δίνεται δυστυχώς να παραστεί σήμερα επειδή γνωρίζετε το πρόβλημα του Ισλανδικού ηφαιστείου, δεν μπορεί να ταξιδέψει λοιπόν. Θα ήθελα να κάνω ίδιο στην παρουσία των εργασιών που διεξήχθησαν και τα αποτελέσματα που πέτυχε κανείς εκεί και αυτό να το προσπαθήσω να το κάνω σε λίγα λεπτά εγκρίθηκε, σας το λέω με χάρα, ή μάλλον να διορθώσω, επετέφθη ακριβώς ε, στον τρίλογο αυτό μια συμφωνία σχετικά με την θεώρηση του κανισμού για ορισμένα ειδικά μέτρα υπέρ τις ε, υπερπεριφερειακές ε, γεωργικές περιοχές. Βρέθηκε, επετεύχθη αυτός ο συντονισμός, αυτή η συμβαστική λύση με την Ισπανική Προεδρία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω. Αυτή η συμβαστική λύση συμπεριλαμβάνει ανταποκρίνεται στα κύρια τα οποία έχουμε ζητήσει εμείς εδώ στην Επιτροπή μας και ειδικότερα σε μια εξαίρεση ώστε στις Αζόρες να μπορέσουν να αναδιαρθρώσουν τη βιομηχανία τους ακριβώς επειδή δεν θα ισχύουν οι ποσοστώσεις γάλακτος άρα λοιπόν με κατάλληλη προσαρμογή της παραγωγής και επίσης μόνιμη εξαίρεση ώστε τα Κανάρια νησιά να μπορούν να συνεχίσουν να προμηθεύονται με φυτικό λίπος ε, σκόνη σε γάλα. Και την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ακριβώς ε, για να μπορέσουν να ισχύσουν όλα αυτά όσο γίνεται συντομότερα θα υπάρξει μια συνάντηση και να ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2010. Θα κατεθεί λοιπόν ο φάκελος αυτός εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων υπομορφή μιας ε, τροπολογίας που έχει, θα ενσωματωθεί στην έκθεση Αλντες για τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι έχουν συνυπογράψει αυτή την τροπολογία που θα ενσωματωθεί ότι η προθεσμία ορίστηκε για την Τετάρτη την επόμενη στις 12 του μήνα το αργότερο για την κατάθεση τροπολογιών και για τη γραμματεία. Ακριβώς για την κατάθεση αυτή για την Ολομέλεια έχουμε την Τετάρτη στις 12 Μέχρι τότε είναι η προθεσμία. Εξ ονόματο τη Επιτροπή μα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μα και όλη την ομάδα των διαπραγματευτών και να ευχαριστήσω και του συναδέλφου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου που μα επέτρεψαν έτσι επιτυχώ να έχουμε, να ολοκληρώσουμε σε συναπόφαση την πρώτη έκθεση μετά από την θέση ισχύ τη Συνθήκη Λισαβόνα. Αν δεν έχετε να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, υιοθετείτε έτσι η μεσιά διάταξη και αν κανείς δεν επιθυμεί το λόγο μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ομάδα εργασίας μας. Αυτά. Έχουμε σε web stream άμεση αναμετάδοση της σημερινής συνάντησης. Ε, η υπουργό Έλενα Εσπινόζα θα έλθει σε λίγο εδώ. Μας είχε ενημερώσει ότι θα καθυστερήσει λίγα λεπτά. Θα έρθει σε λίγο λοιπόν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα-δύο λεπτά μια κάποια παρουσίαση θα σας κάνω και μετά το λόγο θα έχει ο Ντάσιαν ο Επίτροπος το λόγο θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ και δείχνει έτσι την διάθεσή του να συνεργαστεί με την Επιτροπή μας. Ξεκινάμε λοιπόν ε, αυτή την ομάδα εργασία ε, για την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού μας συστήματος που είναι ουσιώδες σημείο για το μέλλον ε, των γεωργών μας και των εργοτικών περιοχών μας για την προοπτική αυτή, αυτές οι ρυθμίσεις εμπορικές είναι από τα κύρια σημεία πάνω στα οποία πρέπει να εργαστεί κανείς. Δεν είναι τυχαίο που ήταν από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας από όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της όπως η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου Εσπινόζα αρκετές φορές το επανέλαβε με τη σημερινή ομάδα εργασία θέλουμε στην Επιτροπή μας να μπορέσουμε να συλλογιστούμε και να βαθύνουμε πάνω στο θέμα αυτό και να μπορέσουμε να αποφεληθούμε από την παρέμβαση εμπειρογνωμόνων και με τη συμμετοχή και με την Προεδρεύουσα Εσπινόλιζα και με τον Επίτροπο Ντάσιον Σιόλος, τον οποίο ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Αυτό που συζητάμε έχει ιδιαίτερη σημασία για να εγγυηθούμε ότι οι προσπάθειες ευρωπαϊκές στην ποιότητα, στην ευμάρεια των ζώων, στην υγιεινή διατροφή να μην είναι κάτι το επειδή η αγορά θα είναι ανίκονη να αναγνωρίσει τις ε, κοινωνικές αξίες ε, που πάνε μαζί με το ίδιο το προϊόν. Ε, θα πρέπει να προσέχουμε τις επιπτώσεις από τη διαστρέβλωση που προκαλούν όσοι δεν υπόκεινται σε αυτό και ευνοούνται έτσι ανταγωνιστικά ε, ακριβώς και αυτό και για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού μας συστήματος και να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό σύστημα και μαζί και τις εγγυήσει και τόσα ισχύουν για τους καταναλωτές πολίτες μας. Από τις κύριες προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε είναι η προώθηση μιας αγοράς περισσότερο διάφανης ε, και που θα προσανατολίζεται στην προμαζόμενη αμοιβαιότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος για ε, να μπορέσουμε έτσι να αντισταθμίσουμε την αδυναμία της αγοράς, να αναγνωρίσει αυτές τις κοινωνικές αξίες προϊόν και επίσης μια μεγαλύτερη σύγκληση σε διεθνές επίπεδο των προτύπων των κοινωνικών περιβαλλοντικών για να αποφύγουμε ώστε αυτά τα πρότυπα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να είναι όχι μια ευκαιρία για τους καταναλωτές μας αλλά αντίθετα είναι κάτι το επιβλαβές για τους γεωργού μας θα πρέπει να καταλάβουμε το βέλτιστο δρόμο για να προσεγγίσουμε περισσότερο και επαρκώς αυτή την προοπτική. Ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι δεσμοί διαπραγματευτικοί και ποιες είναι οι δυνατότητες για να επισπιστούμε ένα πρότυπο για τους πολίτες μας μετά από την εισαγωγή της εργασιών που θα ζητήσω από την ε, μετά από τον Επίτροπο Ντάσιαν Σιόλος θα ζητήσω ακριβώς να λάβει το λόγο η Σπινόζα τρεις εμπειρογνώμονες. Ε, ο Χωσέ Μαρία Εσπούνη από την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή που θα μας μιλήσει για την ανάγκη να ενισχύσουμε το αγροτροφικό διατροφικό πρότυπο το ευρωπαϊκό. Επίσης η κυρία Μαρία Άντζελα Παρίτ από αγρονόμο από την ΙΝΕΑ που θα μας μιλήσει για όλες αυτές τις υποχρεώσεις διοικητικές και τις ρυθμίσεις κοινοτικές μαζί με το πλαίσιο του διεθνές το εμπορικό για τον γεωργικό τομέα και θα έχουμε και τον Αμπτελ Χακίμ Χαμούντι από το ΙΝΡΑ που είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονομικών Ερευνών που θα μας μιλήσει για τις υποχρεώσεις διοικητικές και τις ρυθμίσεις κοινοτικές για τον γεωργικό τομέα και πώς επηρεάζουν όλα αυτά την αγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Όπως συνήθως δε, μετά από την παρέμβαση των εμπειρογνωμών θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με δικές σας ερωτήσεις και λοιπά και παρεμβάσεις. Μία ώρα και 15 λεπτά στο σύνολό τους. Ευχαριστούμε όλους και δίνω το λόγο αμέσως στον Επίτροπο για να κάνει την εισαγωγή του θέματος. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος λοιπόν. Paolo. Ευχαριστώ Παύλο. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να με βλέπετε γιατί σε ένδειξη βασμού προς το κοινοβούλιο πήρε μια καρέκλα που είναι χαμηλότερη αυτή του Προέδρου. Αλλά δεν θα με εμποδίσει αυτό να συζητήσω με και την ουσία του θέματος, πράγματα άλλωστε τα οποία έχουμε δει και όταν συστήσαμε το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα και την διαφύλαξη του ε, γεωργικού προτύπου της Ευρώπης, του γεωργικού μοντέλου της Ευρώπης. Και νομίζω ότι, όπως άλλωστε είπε και ο Πρόεδρο, ότι αυτό είναι το κεντρικό αντικείμενο της συζήτηση σήμερα. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα διατηρήσει και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, χωρίς ωστόσο να απολέσει τα χαρακτηριστικά της εκείνα στοιχεία που την κάνουν ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη στις παγκόσμιες αγορές. Και όχι μόνο βέβαια ε, στο εξωτερικό αλλά και εδώ στην ευρωπαϊκή αγορά. Έκαναν λοιπόν ε, οι διοργανωτές αυτής της συνάντησης ε, το συσχετισμό μεταξύ της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των κανόνων δηλαδή των προδιαγραφών και της ανταγωνιστικότητας. Και θα ήθελα ξεκινώντας να επισημάνω ότι αυτές οι προδιαγραφές που καλούνται να σέβονται οι παραγωγή μας με τα ε, προϊόντα τους είναι αυτές οι προδιαγραφές τις οποίες έχει μάθει που γνωρίζει από τα διατροφικά προϊόντα ο πολίτης, ο καταναλωτής. Όταν Δηλαδή εξασφαλίστηκε η αυτάρκεια μας, οι επαρκείς ποσότητες στις αγορές μας και μπορέσαμε να προχωρήσουμε προς μια πιο αυστηρή επιλογή ποιότητας και ως προς την ε, γεύση αλλά και ως προς την ποιότητα παραγωγής όχι δηλαδή μόνο στο αποτέλεσμα του ελληνικού γεωργικού προϊόντος αλλά και ως προς τον τρόπο παραγωγής γιατί έχουμε και εδώ προδιαγραφές για τον τρόπο παραγωγής για τις επιπτώσεις ενδεχομένως των περιβάλλον ή την ευημερία των ζώων και ως εκ τούτου με τον τρόπο αυτό σταδιακά οικοδομήθηκε το ευρωπαϊκό πρότυπο ε, αγροτικών προϊόντων διατροφής που είναι γνωστό όλο και περισσότερο στις διεθνείς αγορές, γιατί και τα προϊόντα μας είναι όλο και πιο ε, παρόντα στις διεθνείς αγορές, αλλά ταυτόχρονα και γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχουμε όλο και πιο εντατικές ε, διαπραγματεύσεις πολυμερής μέσα από το γύρο της Δόχα στον ε, οποίο, στο πλαίσιο του οποίου συζητούνται θέματα αγροτικών προϊόντων διατροφής. Και έτσι θα πρέπει να ε, διερωτηθούμε συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό αγροτικό προϊόν διατροφής, το οποίο έχει ε, παραχθεί με βάση και την επιθυμία και τις προτιμήσεις του καταναλωτή και φορολογουμένου της Ευρώπης θα μπορέσει να διατηρηθεί, θα εξακολουθεί να παράγεται χωρίς όμως να βρεθούν σε μειονέκτημα ανταγωνιστικό η γεωργή μας, η παραγωγή μας από την άλλη πλευρά. Υπογραμμίζω λοιπόν αυτή τη διάσταση διότι πρέπει αυτές οι προδιαγραφές να αναγνωρίσουμε ότι είναι απόρρια των ε, επιλογών, των προτιμήσεων του φορολογούμενου Παύλα καταναλωτή και το πώς θα τηρηθούν αυτές, εάν ενδεχομένω θεωρεί κανείς ότι η έλεγχη είναι υπερβολικά γραφειοκρατική, οι διαδικασίες για την αναγνώριση των προδιαγραφών είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές. Το πρόβλημα της γραφειοκρατίας είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική τρόπον την ε, αντίληψη, η επίκριση. Ε, στη συνέχεια έχουμε βέβαια να δούμε και τον καταναλωτή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διάκριση που έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων, food safety, προδιαγραφές δηλαδή μη διαπραγματεύσιμες, δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε ούτε με τους διεθνείς μας εταίρους, γιατί έχει να κάνει όχι μόνο με την ποιότητα των προϊόντων, αλλά με την ίδια τη δημόσια υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Και έτσι η προϋπόθεση αυτή αποτελεί στοιχείο συστατικό του ορισμού του ευρωπαϊκού προτύπου προϊόντων, γεωργικών προϊόντων διατροφής. Έτσι λοιπόν η φυτοϊγειονομική που ξέρετε δεν ανήκει στο δικό μου ε, πεδίο δραστηριοτήτων γιατί είναι ζήτημα δημόσιας υγείας ε, αλλά πάντως δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ούτε, μέσα στο, ούτε με τους διεθνείς μας εταίρους και πολλές φορές όπως γνωρίζετε εμποδίσαμε την εισρωή στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων που δεν σέβονταν τις προδιαγραφές ε, δημόσιας υγείας και υγιεινής των τροφίμων, ασφάλειας των τροφίμων. Η Επιτροπή ήταν πάντοτε άτεκτη σε αυτό το θέμα και σας διαβεβαιώ ότι θα εξακολουθήσει να παραμένει άτεκτη. Επίσης, έχουμε να κάνουμε με προδιαγραφές που απορρέουν από τις ειδικέ ευρωπαϊκές, ιδιαίτερε αν θέλετε, ευρωπαϊκές προτιμήσεις, δηλαδή και την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, προδιαγραφές ποιότητας εν προκειμένου, που διαφοροποιούν τα προϊόντα το ένα από το άλλο. Και σε τι αυτή περίπτωση οι προδιαγραφές απορρέουν Μένω, όπως είπαμε, από μια ιδιαίτερη προτίμηση από την ευρωπαϊκή αγορά και τις έχουμε ως εκ τούτου ε, προστατεύσει, τις έχουμε εισαγάγει μέσα σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και μπορούμε να τις προστατεύουμε μόνο μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά απόλυτα, χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να τις επιβάλλουμε αυτές καθεαυτές στους διεθνείς εμπορικούς μας εταίρους ή τουλάχιστον δεν μπορούμε αυτόματα να τις επιβάλλουμε. Και δι' αυτό θα πρέπει ορισμένα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη και για το μέλλον δεν ε, μπορούμε βεβαίως να ε, υποχωρήσουμε ως προς τις απαιτήσεις μας. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τις απαιτήσει ποιότητας. Θα πρέπει αντιθέτως πιστεύω να τις αναβαθμίσουμε κατά τρόπο να αντιληφθούν και οι εταίροι μας ότι δεν πρόκειται για ε, μη φραγμού ή για τεχνητούς φραγμούς ω προ την είσοδο ενό προϊόντος στην αγορά, αλλά ότι έχουν να κάνουν με, την, ε, με τις αξίες μας, με τις απαιτήσει και, προ, και προτιμήσεις των καταναλωτών, αλλά και με την αξία που, έχει, που, που σημαίνει σεβασμός της ευημερία των ζώων, σεβασμός μιας βιώσιμης αηφόρου γεωργίας κτλ. Και ίσω εν προκειμένου θα έπρεπε να βελτιωθεί η διεθνή διακυβέρνηση στο θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε, να βοηθήσουμε μάλλον στην ανάπτυξη διεθνών ε, διαγραφών ε, στο πλαίσιο και του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, στο πλαίσιο του Κόντεξ Αλιμεντάριους. Και πρέπει να επισημάνω ότι είχαμε μια συζήτηση προ ανατολισμό στο πλαίσιο της Επιτροπής ως λογικού οργάνου για τις διεθνείς διαπραγματεύσει. Μια συζήτηση από την οποία προέκυψε πως συμφωνούμε να υποστηρίξουμε μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσει και την προαγωγή των δικών μας προδιαγραφών ω αξιών που απαιτούμε να γίνονται σεβασμές προκειμένου να εξασφαλιστεί αεφόρος γεωργία όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί αυτό, ξέρω ότι δεν είναι και μόνη λύση για να φτάσουμε στον ίδιο στόχο, αλλά πάντως θα συνεχίσουμε με αυτή την προσπάθεια όσο μπορούμε. Και όσο περνάει από το χέρι μου, εγώ θα επαγρυπνώ για αυτό το στόχο. Και άλλοι επιτροποί, επίση σα διαβεβαιώ, σε άλλα χαρακτηροφυλάκια συναφή, έχουν επίση δεσμευθεί και έχουν την ίδια άποψη Εν συνεχεία, πρέπει να δούμε με ποιο σύστημα στήριξη στη γεωργία προσαρμοσμένο στις συνθήκες από το 2013 και μετά θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε και να αναβαθμίσουμε τον σεβασμό αυτών, την τήρηση αυτών των προδιαγραφών γιατί πολλές φορές οι προδιαγραφές αυτές ε, γίνονται, ε, ε, αναγνωρίζονται ω προδιαγραφές προστασία ενό δημόσιου αγαθού, γιατί ω τέτοιο αντιλαμβάνεται τα προϊόντα διατροφής, τα γεωργικά προϊόντα διατροφή ο καταναλωτής. Άρα πρέπει ω τέτοια και εμεί να τα προστατεύσουμε από τι προδιαγραφές μας και να βρούμε κατάλληλε προδιαγραφές για τέτοιου είδου προϊόντα. Ε, τρίτον, δε, πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τον παραγωγό να κοινοποιεί καλύτερα, να ενημερώνει καλύτερα, να προβάλλει καλύτερα την υπεραξία του προϊόντος του, αυτή, την οποία, ε, αυτή η οποία ενδεχομένω υποκρύπτεται πίσω από ένα όνομα, πίσω από μια προέλευση, δηλαδή προδιαγραφές ποιότητας, προδιαγραφές ε, ποικιλία επίση των προϊόντων μα, των γεωργικών μα προϊόντων διατροφή, που εάν την αξιοποιήσουμε με τρόπο ευφύ μπορούμε να την ε, καταστήσουμε ιδιαίτερο πλούτο και κέρδο για την γεωργία μα. Η διαφοροποίηση δηλαδή, με βάση βέβαια όχι κάποια τυχαία επιλογή, αλλά ε, με βάση τα προϊόντα, την προέλευσή τους και τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά, θα πρέπει να προβληθεί ώστε και να γνωρίζει και να αναγνωρίζει όταν αγοράζει ένα προϊόν ο καταναλωτής και θα είναι ο τρόπος να εξάρουμε και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις προσπάθειες του παραγωγού για την παραγωγή του πρόοδος αυτού. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία ενός νομοθετικού, μιας δέσμης νομοθετικών μέτρων για τα προϊόντα ποιότητας, τα τρόφιμα ποιότητας που έχει υποβληθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει εξεταστεί μέσα από την έκθεση Σκότα, έχει λάβει τις απαντήσεις, η πρόταση της Επιτροπής, οποίε βεβαίω θα λάβουμε υπόψη, τις απαντήσεις που δίνει αυτή η έκθεση. Θα τη συζητήσουμε και στην Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη επίση έτσι ώστε να δώσουμε ακριβώ την έμφαση σε αυτό που είπα, την ποιότητα, τη διαφοροποίηση των προϊόντων, έτσι ώστε να έχουμε το ευρύτερο δυνατό φάσμα ως προσφορά ε, γεωργικών προϊόντων διατροφής για τον καταναλωτή μας και κατά τρόπον αναγνωρίσιμο και αναγνώσιμο για τον καταναλωτή. Όχι μόνο δηλαδή γεωγραφία, ε, όχι μόνο ε, ονομασία γεωγραφικής προέλευσης ή ονομασία προέλευσης ή διαφορετικές ή ιδιωτικές εντός εισαγωγικών ε, προδιαγραφές ποιότητας, αλλά και ένα μηχανισμό ο οποίος θα μπορεί να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα και χαρακτηριστικά κάποιες περιοχής προϊόντα. Φέρει πίν της ορεινής κτηνοτροφίας ή διαφόρων περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα είδαμε και με την έκθεσή σα, την έκθεση του Κοινοβουλίου, όπω είπα και νωρίτερα. Πάντω θέλουμε πάνω απ' όλα να αναδείξουμε τι προσπάθειε των ε, παραγωγών μα. Τούτου λέχθόντο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει και να απορρίπτουμε κάθε έννοια ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Αλλά θα πρέπει να αναπτύξουμε μια στρατηγική ώστε αυτέ οι διεθνεί συναλλαγές να επιτρέπουν καλύτερη αναγνώριση των προϊόντων μας. Οι συζητήσεις σας σήμερα ίσως να προβάλλουν και άλλες πτυχές τις οποίες δεχομένως παρέλειψα στην παρουσίασή μου. Σας διαβεβαιώνω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω και θα ακούσω οποιαδήποτε πρόταση είναι σχετική με το πακέτο και τη διαφοροποίηση των προϊόντων και βέβαια τις, ε, τους μηχανισμούς που θα θεσπίσουμε για την κοινή γεωργική πολιτική από το 2013 και έπειτα. Έτσι ώστε και να διαφυλάξουμε τις γεωργίες μας, τις γεωργικές μας παραγωγές, την, διαφορε... την ιδιαιτερότητα δηλαδή της γεωργικής παραγωγής σε κάθε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε και ο παραγωγός να είναι σε θέση να βλέπει ότι η ε, γεωργική παραγωγή, όπως την προάγουμε, όπως την επιδιώκουμε, λαμβάνει υπόψη και τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις και όχι μόνο τις προτιμήσεις της αγοράς, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, θα θέλω να το υπογραμμίσω. Θέλουμε μια κοινή γεωργική πολιτική στο μέλλον η οποία θα ικανοποιεί τις προσδοκίες κάθε πλευράς, όχι μόνο τις ανάγκες της ποιότητας ή της ποσότητας που θα ειστρέψει στην αγορά, αλλά και όλων των παραγόντων που ε, μετέχουν στην γεωργία. Βέβαια, μερικέ φορές είναι εύκολο να λέμε ότι θα ε, διαλύσουμε κάποιο προηγούμενο σύστημα γιατί διαπιστώνουμε ότι δεν είναι ικανοποιητικό και δεν ε, ε, φέρνει αποτελέσματα ή να αγνοήσουμε τις προσδοκίες κάποιων γιατί είναι πολύ δύσκολο να τις ικανοποιήσουμε όμως εμείς θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε να προχωρήσουμε σε ικανοποίηση τελικά όλων αυτών των προσδοκιών και επιθυμιών. Και κλείνοντα, θα ήθελα να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά τη διάκριση μεταξύ των προδιαγραφών και τη εφαρμογή αυτών. Στην εφαρμογή των προδιαγραφών, ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να απλουστευτεί κυρίω το γεωγραφικό βάρος, αλλά πάντως θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο ε, φιλοδοξιών υψηλό σε σχέση με αυτές τις προδιαγραφές διότι έχουν κάποιο λόγο που υπάρχουν στις κοινωνίες μας, προσφέρουν κάτι στις κοινωνίες μας και εφόσον προσφέρουν κάτι το θετικό στις μας πρέπει οπωσδήποτε να τι λαμβάνουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής σα ε, για την συζήτηση αυτή. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη και στο Συμβούλιο και άρα θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για ε, έξεφραση απόψεων ε, και συναγωγή συμπερασμάτων. Θα παρακολουθήσουμε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. σα ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Επίτροπε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω και για όσα τόνισες και ότι είπες ότι είσαι διαθέσιμος, ε, ακριβώς έχεις διάθεση να τονίσεις ε, αυτά τα στοιχεία και με αυτή την έκθεση σκοτά για το θέμα της ποιότητας και έτσι ορισμένες προτάσεις μας να μπορέσουν να υιοθετηθούν, να σωματωθούν στην νομοθετική πρόταση την οποία συντάσσει, θα συντάξει για το φθινόπωρο μας έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ξεκινήσω αμέσως ε, δίνοντας το λόγο στους εμπειρογνώμονες μας. Ε, μόλις με πληροφόρησαν ότι η Υπουργός Εσπινόσα θα φτάσει σε λίγο. Ζωζέ Μαρία Εσπινή που θα μας μιλήσει για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού ευρωπαϊκού προτύπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την πρόσκληση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για να σας παρουσιάσουμε την έκθεσή μας για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μοντέλου παραγωγής γεωργικών προϊόντων διατροφής. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η ΟΚΕ λειτουργεί με τρεις ομάδες διαφορετικών ε, συμφερόντων, εργαδοτών, εργαζομένων και διαφόρων ε, δραστηριοτήτων. Και αυτή η γνωμοδότηση, αυτή η έκθεση είναι ο καρπός ε, των εργασιών μιας ομάδας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τρεις ομάδες και μάλιστα εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, 128 ψήφους υπέρ, μία ψήφο και τρεις αποχές. Θα πω καταρχήν κάτι αυτονόητο. Η γεωργική πολιτική είναι η πρωταρχική κοινοτική πολιτική και πρέπει να θεωρηθεί ως ε, τομέα στρατηγικής σημασίας. Για μία πεντηκονταετία συνέχισε τις σταδιακές προσαρμογές για να εκπληρώσει τους στόχους του. Καταρχήν εφοδιάσει με τρόφιμα ε, σε μεταπολεμική περίοδο και εποχή σπάνια σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και να εξασφαλίσει τον ανεφοδιασμό σε υγιή και ασφαλή προϊόντα ε, με τις κανονικές κοινωνικο-οικονομικές περιστάσεις και με σεβασμό προς το περιβάλλον. Διατηρώντας λοιπόν μια θετική αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής, όπως κάναμε μέχρι τώρα, ίσως θα πρέπει να επανεξετάσουμε ορισμένα κέρια σημεία της. Μεταξύ αυτών βρίσκεται καταρχήν η ανάγκη εφοδιασμού μας με μηχανισμούς που θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν αυτή τη μεγάλη ρευστότητα και μεταβλητότητα των ε, τιμών πρώτων υλών, τις οποίες γίναμε μάρτυρες και μας τύχησε πάρα πολύ. Επίσης, όπως είπε και ο Επιτροπός, τα θέματα ιδιαιτεροτήτων το τομέα αυτού, γεωργικές ονομασίες προέλευσης, προ, προστατευόμενη γεωργική προέλευση, κάποιες, κάποια παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και υψηλέ τεχνικές προδιαγραφές για να ενισχύσουμε το μοντέλο και να προασπίσουμε καλύτερα το γεωργικό μας μοντέλο στις εξωτερικές αγορές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και γεωργικής προέλευσης που δεν έχουν ε, νόημα ούτε και ουσιαστικό περιεχόμενο. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια πολιτική προώθησης και διαφήμισης της ε, γεωργίας μας ε, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την εμπορική αξία των γεωργικών προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια στρατηγική άποψη για την γεωργοτροφημική αλυσίδα να πατάξουμε τις καταχρηστικές μεθόδους, ε, η κατάχρηση δεσπόζας θέσης ή στρεβλό ανταγωνισμού. Το 2007 καταρτίστηκε μία μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 17 χωρών μελών και είπαμε, είδαμε ότι οι τρεις πρώτοι διανομής σε μία ευρωπαϊκή χώρα κάλυπταν το 80% των άμεσων ε, πωλήσεων. Σε άλλη 75%, σε τρεις χώρες πάνω από 60% και σε άλλες έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση ήταν πάνω από 50% η μεγαλοδιανομή. Επίσης, σε 10 χώρε ο πρώτος διανομέας υλοποιεί πάνω, το 20, από, το, πάνω από τα 20% των άμεσων ε, πωλήσεων. Είναι χαρακτηριστικά αυτά τα στοιχεία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επιπλέον, διαπιστώνουμε, σε ό,τι αφορά ε, τους σε ορισμένε η μάρκα είναι σημαντική και, και το, εμπορικό σήμα και αντιπροσωπεύει 40% σε ορισμένε χώρε, 35% των πωλήσεων σε άλλε χώρε. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η συγκέντρωση γίνεται όλο και μεγαλύτερη και είναι όλο και πιο σαφή η συγκέντρωση των πωλήσεων στι ε, μεγάλε αλυσίδε παραγωγή. Ε, διανομή, συγγνώμη. Γι' αυτό, όπω είπε και ο Επίτροπο, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ενημέρωση προ τον καταναλωτή και φυσικά να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε και τι νέε τεχνολογίε πληροφορία. Είναι σαφές ότι το σύστημα αυτό το αγοραπιστιστικό έχει δικές του ανάγκες και θα πρέπει αυτές οι ανάγκες να ληφθούν υπόψη στη νέα γεωργική πολιτική. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε έναν ισχυρό και ανεξάρτητο στρατηγικό τομέα όπως είναι η γεωργία. Το γεωργοτροφημικό μας σύστημα στηρίζεται στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αηφορία και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια στοιχεία όπως την ενίσχυση της ε, ανιχνευσιμότητας, της συχνηλεσιμότητας, της ασφάλειας των προϊόντων, την εφαρμογή πρακτικών που θα σέβονται τον περιβάλλον όπως ολοκληρωμένη παραγωγή, η εφαρμογή κάποιων διατάξεων για την ευημερία των ζώων, η λήψη υπόψη κοινωνικών ε, διατάξεων όπως της προστασίας των εργαζομένων και όλα αυτά ενισχύοντας ταυτόχρονα την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τις γεωργικές μας παραγωγές και να ανταποκριθούμε στη μείζωνα πρόκληση της προσπάθειας ξερίζωσης του λοιμού, την πείνα στον κόσμο. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν τεράστιες προσπάθειες και διαπιστώσαμε πολύ σημαντικά κενά. Κενά και αδυναμίες που θα πρέπει να τα εντοπίσουμε για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Για παράδειγμα, νευραλικό σημείο είναι το θέμα της εισαγωγής των τροφίμων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο πρώτος εξαγωγέας και ο πρώτος εισαγωγέας παγκοσμίω. Παρ' όλα αυτά, ο νομοθέτης ήταν πολύ αυστηρός για την ε, κοινοτική παραγωγή και άφησε σε δεύτερη μοίρα τις ε, εισαγωγές από τρίτες χώρες. Εκεί υπάρχει διαφορά μεταχείριση ό,τι αφορά την εχληνασιμότητα μεταξύ των κοινοτικών και των έξω κοινοτικών προϊόντων. Στα κοινοτικά προϊόντα η χνηλασιμότητα καλύπτει όλη την αλυσίδα, από το χωράφι μέχρι το τραπέζι. Ενώ για τα εισαγόμενα προϊόντα είναι από τα σύνορα μέχρι το τραπέζι η χνηλασιμότητα. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την εχνηλασιμότητα σε προϊόντα τρίτων χωρών που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα κοινοτικά προϊόντα. Για παράδειγμα, το θέμα της ευημερίας των ζώων. Μερικές φορές μάλιστα, τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες χαίρουν ε, προνομιακής ε, δασμολογική μεταχείρισης. Και δεν είναι ίσονο σημασία ε, ότι ένα τρίτο των καταγγελιών που γίνονται για τρόφιμα αφορούν εισαγόμενα προϊόντα. Επίσης, το ρυθμιστικό κόστος για την κτηνοτροφία, για παράδειγμα, ή τη χρήση κτηνοτροφικών προϊόντων. Εκεί μας λείπουν πρώτες ύλε. Και ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν σαφείς περιορισμοί σε ό,τι αφορά τη χρήση ε, προϊόντων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, αντίστοιχη αυστηρή νομοθεσία δεν ισχύει για τα εισαγόμενα προϊόντα, οπότε δεν ε, υλοποιείται στην πράξη ο υψηλό βαθμό προστασία του καταναλωτή, γιατί εισάγονται προϊόντα που περιλαμβάνουν τέτοιου γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού. Στη γνωμοδότηση δεν ταχθήκαμε ούτε υπέρ ούτε κατά των γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών. Αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι η παρούσα κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει ε, τεράστιες απώλειες ε, της τάξης των 200 δις στην αγροεπιστηστική βιομηχανία. Επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε τις πιο εντατικές εργατικό δυναμικό παραγωγές και μάλιστα σε περιοχές που εξαρτώνται πλήρως ή σχεδόν πλήρως από μία και μόνο καλλιέργεια. Και η βιομηχανία που καλύπτει τέτοιο προϊόν, τέτοια, γεωρική παραγωγή, θα πρέπει επίση να προστατεύεται. Δεν είναι λογικό λοιπόν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί να υφίστανται δυσμενή μεταχείριση στη φυσική του αγορά έναντι τρίτων εξοκοινοτικών. Και μάλιστα αυτή η διακριτική μεταχείριση να πηγάζει από την ίδια την κοινοτική νομοθεσία. Κατά τη γνώμη τη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσει και σε ορισμένε περιπτώσει θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτές σταδιακά και προοδευτικά. Για παράδειγμα, θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης στην αγορά, να γίνεται καλύτερος έλεγχος των εισαγωγών, ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα κοινοτικά προϊόντα και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για τους ε, καταναλωτές. Θα πρέπει να εξαγάγουμε το γεωργικό μας μοντέλο και να προωθήσουμε την εναρμόνιση και των υπόλοιπων νομοθεσιών με τη δική μας να προωθήσουμε την αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων ε, ευημερία ζώνη προστασία των καταναλωτών με τι τρίτε χώρε και να περιλάβουμε τέτοιε ρήτρε στα ειδικά κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών για την ε, αμοιβαία αναγνώριση συστήματο σε θέματα υγειονομικά, φυτογειονομικά και διατροφικά. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την παγκόσμια τεχνική αρρωγή. Να συνεργαστούμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι εξαγωγή ή δυνάμει εξαγωγής ε, πρώτων υλών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην κατάρτιση, καλύτερη κατάρτιση των τεχνικών, την εκπόνηση ποιοτικών προδιαγραφών και την ανταλλαγή υπαλλήλων. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε εμπορικά χρηματοπιστωτικά κίνητρα και κίνητρα συνεργασίας αναπτυξιακής προ τι χώρε που εναρμονίζουν το σύστημά του με το κοινοτικό σύστημα. Επιπλέον θα πρέπει να βελτιώσουμε την ομοθεσία μα. Όπως είπε και ο Επίτροπο θα πρέπει να περιορίσουμε το γραφειοκρατικό άχθο που μερικέ φορέ εμποδίζει την εύρυθμη ανάπτυξη τη βιομηχανία. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, όχι από το γεωργικό τομέα. Ε, συνέταξα μία γραμμοδότηση και για την υδατοκαλλιέργεια και διαπίστωσα ότι σε ορισμένε χώρε την τελευταία 15 ετία δεν εγκρίθηκε ούτε μία άδεια για την κατασκευή ε, καταστάσεων υδατοκαλλιέργεια. Πώ είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά μα με τέτοια κολλησιέργεια. Επίση θα πρέπει να θεσπίσουμε συστήματα που να εμποδίζουν τη μετεκατάσταση επιχειρήσεων προς άλλες ζώνες με χαμηλότερο μισθολογικό κόστος και ίσονο σημασία κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να προωθήσουμε κανόνες αξιοπρεπούς εργασίες και να, περιλα... να τις περιλάβουμε ως ρήτρε στις εμπορικές μας συμφωνίες. Επιπλέον πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ε, αποκατάσταση της ισορροπίας. Και να σας δώσω και κάποια στοιχεία για την ε, βιομηχανία παραγωγή γεωργικών προϊόντων. 965 δι είναι ο τζίρο. 310.000 είναι οι επιχειρήσει, πάνω από 99% αυτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσει. 58 δις εκατομμύρια εξαγάγουμε και 57 δις εκατομμύρια εισάγουμε σε γεωργικά προϊόντα. Και μάλιστα, αν το 2009 αντιπροσωπεύαμε το 17,5% των διεθνών συναλλαγών, το 98 ήμασταν το 24,6%, Το 24,6%. Δηλαδή χάνουμε με τα χρόνια την ανταγωνιστικότητά μας. Και μάλιστα έχουμε 4.400.000 εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο και μάλιστα παράγουν πολύ περισσότερες θέσεις επασχόλησης από ό,τι χημική βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χωσέ Μαρία Εσπούνη για την εισηγήσή του. Η Προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυρία Εσπινόζα, μόλις αφήχθη, θα ήθελα να τη χαιρετήσω. Αγαπητή Έλενα, ξεκινήσαμε μόλις ε, την ε, συνάντησή μας και την ομάδα αυτή εργασίας και να τονίσω θα ήθελα μετά από όσα είπε και ο Επίτροπος την σημασία που αποδίδει η ε, Ισπανική Προεδρία και μόλις ο κύριος Εσπούνη μας είπε πως έχει κατάσταση και ότι υπάρχουν στοιχεία που δημιουργούν ανταγωνιστικές δυσκολίες απέναντι σε άλλους εξαγωγείς από άλλα μέρη του κόσμου που δεν σέβονται τα υψηλά μας πρότυπα τα οποία εμείς σεβόμαστε και τα οποία έχουμε επιβάλει στους παραγωγούς μας και τα οποία στάνταρτς είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε λοιπόν πολλά και διάφορα τα οποία μας απασχολούν και θα ήθελα να λάβεις το λόγο αγαπητή Έλενα και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι δύο. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για την καθυστερημένη μου άφηξη σε αυτή την ακρόαση, σε αυτό το σεμινάριο, αλλά έχουμε όλη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με τις ε, αεροπορικές μεταφορές και ε, τον έφος της ηφαιστιακής τέφρας που μας ήρθε από την Ισλανδία. Θα ήθελα να πω καταρχήν, μπαίνοντα στο κύριο θέμα, ότι οι Ευρωπαίοι έχουμε πολλούς λόγους για να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα τρόφιμά μας. Ενισχυμένοι μάλιστα από την κοινή γεωργική πολιτική, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι προσάρμοσαν τις παραγωγές τους στις ε, εξελίξεις της κοινωνίας μας, ασκώντας τη λειτουργία τους ε, Παρέχοντα τρόφιμα προς τον κοινοτικό πληθυσμό που όλο και αυξανόταν. Στην πορεία μάλιστα αντιμετώπισαν μείζονε προκλήσεις, περνώντας από μια λειτουργία απλού ανεφοδιασμού σε τρόφιμα των κοινοτικών αγορών σε μια πραγματική έφεση ανταγωνισμού στις παγκόσμιε αγορές με μια δική του ταυτότητα που συνάδει με τον πολιτισμό και τις κοινοτικές αξίες. Στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο η γεωργική και κτηνατροφική δραστηριότητα εμφανίζονται όλο και περισσότερο ως στοιχεία που διαμορφώνουν το τοπίο και την ύπεθρο και προσθέτουν στη λειτουργία της παροχής και αναφοδιασμού σε τρόφιμα και άλλα στοιχεία με τη μορφή παροχής περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολιτιστικών υπηρεσιών πρώτης τάξεως. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν το 50% της επικράτειάς μας με άμεση θέση απασχόληση στη γεωργική και αγροεπιστηστική παραγωγή 18,6 εκατομμυρίων ανθρώπων ή αν το προτιμάτε με ποσοστά το 8,6% της συνολικής απασχόλησης στην, στην Ευρώπη. Επιπλέον, η δραστηριότητα της βιομηχανίας παραγωγής γεωργικών προϊόντων διατροφής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του δευτερογενούς ευρωπαϊκού τομέα και περάσαμε από την απλή μεταποίηση στην, στον προσανατολισμό της βιομηχανικής διαδικασίας προς την αύξηση της αξίας των παραγωγών μας. Και μάλιστα η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε ιδιαίτερα στις σταδιακές μεταρρυθμίσεις της κοινή γεωρικής πολιτικής που καθόρισαν τον προσανατολισμό αυτού του αγορεπιστικού κλάδου όχι μόνο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς. Απόδειξη του ανοίγματο αυτού είναι τα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται σε δύο σκέλη με διπλή ιδιότητα και είναι ταυτόχρονα και ο πρώτος εξαγωγές, αλλά και ο πρώτος εισαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής. Ο τομέας αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το 4% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφέ. Το μοντέλο μας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσει ε, και τις αξιώσει των Ευρωπαίων πολιτών ή των Ευρωπαίων καταναλωτών. Επιπλέον θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνίζεται όχι μόνο στην εσωτερική αγορά αλλά και στις παγκόσμιες αγορές. Ιδιαίτερα ο ανταγωνισμός ενισχύθηκε εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης αλλά και των διαδικασιών εμπορικού ανοίγματο που πέραν των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει σε διμερές και πολυμερές επίπεδο πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή διαφαίνεται η διασταύρωση του ευρωπαϊκού αγροεπιστηστικού μοντέλου που είναι καλά εδρεωμένο και προσαρμοσμένο σε μη διαπραγματεύσιμες απαιτήσει που όταν εγκρίθηκαν είχαν τεράστιο πολιτικό κόστος. Το νομοθετικό μέτρο μάλιστα διατροφικής ασφάλειας, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα επερήφανοι, κατάφερε να κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη των καταναλωτών μετά τις κρίσεις που βιώσαμε στο παρελθόν. Επιπλέον φαίνεται και η έφηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφοδιάσει την παραγωγή της με τη δική της ταυτότητα που θα είναι διαφοροποιημένη και θα εγγυάται μια απόλυτη αρμονία μεταξύ των προτιμήσεων των καταναλωτών και των δεσμεύσεων των παραγωγών. Όλα αυτά διαμόρφωσαν ένα μοντέλο παραγωγής τροφίμων που είναι άνευ προηγουμένο και μοναδικό στον κόσμο. Μιλάμε για ένα ιδιάζον ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής ε, γεωργικών τροφίμων. Και μάλιστα το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις ε, που θα πρέπει να πληρούν οι παραγωγές μας. Οι κανόνες αυτοί και τα πρότυπα αυτά αφορούν πολλά και διάφορα ζητήματα, φυτογειονομικά, θέματα υγείας των ζώων ή θέματα ποιότητας τροφίμων και ζωοτροφών. Οι εγγύησει αυτέ βέβαια προποθέτουν ένα συμπληρωματικό κόστο, γιατί οι κανόνε του παιχνιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πανομοιότυπε ε, με τους παγκόσμιους κανόνες. Έτσι στην πράξη ουσιαστικά απαιτούμε παρόμοια, ισοδύναμα τέτοια πρότυπα, ή ισοδύναμες απαιτήσει στις συμφωνίες μας με τις τρίτες χώρες, αλλά εφαρμόζουμε εναρμονισμένα πρότυπα και απαιτήσει στις ενδοκινοτικές συναλλαγές σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής αλυσίδας. Έχουμε διάφορα παραδείγματα υψηλών εναρμονισμένων προδιαγραφών στην Κοινοτική Ένωση, όπως σε θέματα χρήσης ε, παρασιτοκτόνων, θέματα ευημερίας των ζώων, προστασίας του περιβάλλοντος ή την προάσπιση της διαφοροποιημένης ποιότητας ορισμένων τροφίμων. Παρ' όλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι επιτελέσαμε με επιδεξιότητα το έργο μας απέναντι στους διαφόρους παραγωγούς, δυστυχώς δεν καταφέραμε να μεταδώσουμε αυτή την προσπάθεια και τα πλεονεκτήματά της στους καταναλωτές μας. Στο σημείο αυτό λοιπόν ανακύπτει ένα πρόβλημα, γιατί επιβάλαμε μεν μία κοινοτική ρύθμιση στους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς που είναι ανώτεροι των παγκόσμιων κανόνων, αλλά παρόλα αυτά έτσι θέτουμε σε κίνδυνο κάποιους πιο αδύναμους κρίκους της ε, παραγωγικής μας αλυσίδας, όπως είναι οι μικρές βιοτεχνίες ή οι πρωτογενείς παραγωγές που είναι πολύ πιο απομακρυσμένοι από την απόφαση για την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Υπάρχουν λοιπόν ε, εμφανείς αδυναμίες στο παραγωγικό μας μοντέλο και θα πρέπει αυτές να τις αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικό τρόπο και όλα αυτά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να εξακολουθεί να ανεφοδιάζει τις αγορές της και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εξακολουθεί να προσφέρει στους καταναλωτές γεωργικά προϊόντα διατροφής που όχι μόνο είναι ακίνδυνα ή είναι ασφαλή αλλά ταυτόχρονα είναι και ε, ουσιαστικά δημόσια αγαθά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λοιπόν για μερικές προτάσεις δράσεις. Για παράδειγμα, το πρώτο στοιχείο στο οποίο θα μπορούσαμε να δράσουμε, το πρώτο πεδίο, ίσως θα ήταν το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη ρύθμιση που θα βρίσκει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των ανησυχιών του καταναλωτή αλλά και της αηφορίας του παραγωγού οι διάφορες απαιτήσει και προδιαγραφές θα πρέπει να στηρίζονται σε ευρεία κοινωνική συνένεση και να συνοδεύονται από μελέτες επιπτώσεων που θα αξιολογούν ανα πάσα περίπτωση τις ε, οικονομικές συνέπειες όλων των εμπλεκομένων φορέων, όχι μόνο για την εσωτερική αγορά, αλλά και στη διεθνή αγορά, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ισορροπία και να μην δημιουργηθούν ε, περί τη φραγμή στο εμπόριο. Αυτή η επιβεβαίωση λοιπόν της ανάγκης να είμαστε πιστοί στις αρχές ε, του μοντέλου παραγωγής γεωρικών ε, τροφίμων με φέρνει στον επό... στο επόμενο πεδίο δραστηριότητάς μας που είναι η ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών μας για να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο του ευρωπαϊκού παραγωγικού μοντέλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την διαπραγματευτική της θέση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου προσπαθώντας ε, να πετύχει αντίστοιχες απαιτήσει, δίκαιες και αμοιβέ και στους υπόλοιπους οικονομικούς μας εταίρους. Επίσης, η διεθνοποίηση του, των ευρωπαϊκών προδιαγραφών θα, πρέπει, θα πρέπει να ενισχύσουν την εικόνα μας και να βελτιώσουν την πρόσβασή μας ε, στις στρατηγικές ε, παγκόσμιες αγορές και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική μας θέση στον κόσμο οι στρατηγικές ε, προαγωγής των προϊόντων μας στις τρίτες χώρες για να τους ενημερώσουμε για τα πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας είναι απαραίτητη πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλυθεί από κοινού από τους διαφόρους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το ευρωπαϊκό αγροεπιστηστικό μοντέλο θα πρέπει να εκλειφθεί ως ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κυρίως για τους ευρωπαίους καταναλωτές και το δικό του συμφέρον θα πρέπει πρωτίστως να έχουμε κατά νου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τις συλλογικέ μας προσπάθειες για να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με τους καταναλωτές και να τους μεταδώσουμε τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού μας μοντέλου ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν έχοντας καλύτερες γνώσεις και να μπορέσουν να αξιολογήσουν και τα διάφορα προϊόντα. Η ενημέρωση και η κατάρτιση των καταναλωτών θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία της κοινοτικής πολιτικής. Θα πρέπει επιπλέον να διαπιστώσουμε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την προστιθέμενη αξία ενισχύοντας τρεις πυλώνες της εμπορικής ε, αξιοποίησης. Για παράδειγμα, μία απλή ετικετοθεσία που θα είναι ανοιχτή σε όλα τα προϊόντα, εύχρηστη και δεν θα προϋποθέτει σε πληρωματικό κόστος. Δεύτερον, μία γνήσια πληροφόρηση, αληθινή πληροφόρηση του, για το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και των συστημάτων διαφοροποίησης των διαφόρων προϊόντων που περιλαμβάνει. Και τρίτον, μία ισορροπία δυνάμεων στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορευματοποίησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά δικαιολογούνται απόλυτα ακριβώς για τον στόχο να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα αυτού του τομέα στην Ευρώπη και μάλιστα σε κάθε πτυχή, στο σύνολο των αγορών ε, και πέρα από κάθε συγκυρία οικονομική και μάλιστα σε μεμόνιμο τρόπο. Εμείς εργαζόμαστε πάνω σε αρκετές πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν ιδιαίτερα την, ε, για την πληροφόρηση στους καταναλωτές και τις ετικέτες, όπως επίσης ε, και την όλη αλυσίδα αυτών αξιών ε, σε αυτά τα προϊόντα. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν μέσω ενός τρίτου δρόμου και είναι ακριβώς του προσεχούς μοντέλου της Ευρώπης, της κοινή γεωργικής πολιτικής του μέλλοντος. Η Ισπανική Προεδρία έχει ακολουθήσει αυτές τις γραμμές εργασίας όπως το δείχνουν και οι συζητήσεις στα, ε, στα αγροτικά σε αγροτικές συζητήσεις σε επίπεδο συμβουλίου και σίγουρα ε, στηρίζεται και στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οθέτηση αυτών των πρωτοβουλειών. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να συμμετάσχει όλη η κοινωνία σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το θέμα που χρειάζεται μια αμοιβαιότητα σχετικά με αυτά τα προϊόντα. Το σύνολο των στοιχείων είναι σημεία κλειδιά για την οικοδόμηση μιας νέας Ευρώπης και ένας νέος τομέας έτσι που θα πρέπει να ισχύσει για το μέλλον ε, και χωρίς να χάσουμε όμως και τις παλιές βάσεις από τη συνθήκη της Ρώμης μέχρι τη σημερινή συνθήκη της Λισαβόνας και ακριβώς για τον εφοδιασμό των αγορών με ποιοτικά προϊόντα, με λογικές τιμές ε, είναι ένα στόχο που έχει επιτευχθεί από ό,τι φαίνεται, αλλά θα πρέπει να διπλασιάσουμε τι προσπάθειέ μα για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωή σε όλου όσου συμμετέχουν σε αυτήν την αλυσίδα διάθεση προϊόντων, παραγωγής και διάθεση προϊόντων στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ε, μια προσπάθεια και μια ανάληψη υποχρέωση απέναντι στους πολίτες μας. Ε, και εδώ αυτό θα αποτελέσει ένα μοναδικό μοντέλο στον κόσμο και θα μπορέσουμε έτσι και να το δικαιολογήσουμε, να το διατηρήσουμε. Αυτό το πρότυπο είναι η κληρονομιά η δική μας. Θα πρέπει να ενισχυθεί και να διορθεί όπου πρέπει στις διάφορες πτυχές όπου υπάρχουν αδυναμίες και έχουν εμφανιστεί μάλιστα. Εάν δεχτούμε μια μείωση της ανταγωνιστικότητας τότε θέτουμε σε κίνδυνο αυτή την κληρονομιά. Και με την έννοια αυτή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια οικονομία κλίμακα ανώνυμη, χωρίς ανθρώπινο χαρακτήρα. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς το άνοιγμα των αγορών και την πρόκληση αυτή στα πλαίσια μιας διεθνούς φύσεως αυτού του προτύπου του ευρωπαϊκού. Ένας δρόμος υπάρχει μόνο για να πετύχουμε το στόχο μας αυτός ο δρόμος είναι να προσπαθήσουμε όλο είναι περισσότερο στα προϊόντα μας πάνω και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε μία παγίωση ενός ύφου ζωής προτύπου παραγωγής που αφορά όλους μας, έχει να κάνει με όλους μας. Και εδώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, Επιτροπή αυτή τη στιγμή και για την Ισπανική Προεδρία. Θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα για αυτό το στόχο. Θα μπορέσουμε να το πετύχουμε και τα τρία θεσμικά όργανα μαζί μπορούν να το πετύχουν. Αυτό πιστεύω και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την αγαπητή Έλενα. Την ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό και για το πάθος που έδειξε στην εισήγησή της αυτή, για την ενημέρωσή σας και για την ενημέρωση επίσης των καταναλωτών. Αυτά έχουν τρομερή σημασία. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις σε αυτές τις παροτρύνσεις και σε αυτές τις προκλήσεις. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον επόμενο μιλητή, εισηγήτρια μάλλον, την κυρία Μαρία Άντζελο Περίτο από το Γεωπονικό Οικονομικό Ινστιτούτο που θα μας μιλήσει ακριβώς για το θέμα του εμπορικού πλαισίου για τον γεωργικό τομέα. Έχει το λόγο η κυρία Περίτο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Γεια σας σε όλους, είμαι η Μαρία Άντζελα Περίτο, είμαι από το Εθνικό Γεωπονικό Οικονομικό Ινστιτούτο της Ιταλίας, ερευνήτρια και θα ασχοληθώ στην εισήγησή μου στο χάραγμα ενό πλαισίου για το θέμα αυτό και στις απαντήσεις της νομοθετικές και τι ακριβώ γίνεται στο θέμα ε, τα, θέματα τα αγροδιατροφικά είναι περίπλοκα τα θέματα με διάφορες πτυχές θα πρέπει να δούμε από ποια πλευρά θα πρέπει να το εξετάσουμε, πώς θα το προσεγγίσουμε μεθοδολογικά. Εδώ θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην food safety, στην ασφάλεια τροφίμων και το πώς επηρεάζουν όλα αυτά τα πράγματα το παραγωγικό πρότυπο το ευρωπαϊκό και η ποιότητα και η εγγύηση για αυτά τα προϊόντα είναι κάτι που απασχολούν τον πολίτη τον Ευρωπαίο, το ακούσαμε ήδη και θα πρέπει να δούμε και τις απαντήσεις του νομοθέτη του Ευρωπαίου για όλα αυτά τα θέματα. Ήταν συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο 168 ας πούμε κανονισμός του 2002 θα πρέπει να το μια ματιά για να καταλάβουμε ακριβώς ε, τι πλαίσιο χαράσει και θα σας παρουσιάσω τέσσερις διαφορετικές φάσεις το πρώτο μέρος που έχει να κάνει με την μεθοδολογική προσέγγιση για αυτό το food safety που είπαμε, την ασφαλεία τροφίμων και για το διεθνές εμπόριο για το θέμα της ασφαλείας τροφίμων, το πλαίσιο το ευρωπαϊκό για τις καινούριες προκλήσεις και τις μελλοντικές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία στα πλαίσια και των πολύπλευρων ε, συμφωνιών. Οι ανταλλαγές όλες αυτές ε, μετά από τα τελευταία χρόνια ε, μας έκαναν να σκεφτούμε την ποιότητα των προϊόντων, ε, οι καταναλωτές, οι πολίτες και θα πρέπει να πούμε ότι ότι ο καταναλωτής θέλει να είναι υγιεινά τα τρόφιμα, ποιοτικά τα τρόφιμα, ανάλογα βέβαια με τη χώρα με την οποία, από την οποία προέρχεται ο καταναλωτής και ανάλογα με το τι ρυθμίσεις έχει, ε, τι γραμμές έχει χαράξει ο νομοθέτης. Θα πρέπει να δούμε από επιστημονικής πλευράς τι έχει γίνει και με τις διάφορες μελέτες του όσα που λένε ότι ο καταναλωτής δεν έχει στα χέρια του τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνει μια ανάλυση αυτής της ποιότητας ε, και τις, ε, το πόσο εξασφαλίζουν ε, για όλους μας παθογόνους οργανισμούς, καρκινογόνα στοιχεία κλπ. Και δυστυχώς ο καταναλωτής το αντιλαμβάνεται ότι είναι ε, επικίνδυνα αυτά τα προϊόντα μόνο όταν ασθενήσει και μετά. Και όλα αυτά βέβαια προσφέρουν και ένα κίνητρο ε, για να μπορέσουν αυτά τα προϊόντα να είναι υγιεινά, όχι επικίνδυνα, να είναι αθώα σε εισαγωγικά και πολλές φορές ε, βλέπουμε αυτά τα κίνητρα με ειδικά χαρακτηριστικά, με ειδικά πρότυπα Και δυστυχώς όταν ε, αποτυγχάνει η αγορά δεν υπάρχει μια ανταπόκριση, μια αντιστοιχία ανάμεσα σε ζήτηση και σε προσφορά, τότε υπάρχει κάτι το καινούργιο που βλέπουμε με διαφορά, διαφοροποίηση των προτύπων τα οποία ισχύουν πια, με διάφορες πρωτοβουλίες ε, οι οποίες επηρεάζουν τα πράγματα και μάλιστα σημαντικά και που παρεμποδίζουν όμως συχνά και ένα ελεύθερο εμπόριο. Βλέπετε από τη διαφάνεια ακριβώς αριστερά κάτω ότι έχω βάλει ακριβώς όπως το άλμα κοντό βλέπετε τον παραλυσμό που έχω κάνει ο καθένας βάζει τον πύχη σαν κράτος πιο ψηλά, πιο χαμηλά, όπως το επιθυμεί, όπως το πιστεύει. Και η ρύθμιση δε η ευρωπαϊκή τίθεται σε υψηλότερα πάντως σε επίπεδα σχετικά με τον κόντεξ αλιμεντάριος. Θα ήθελα να κάνω και μια μικρή σύντομη παρένθεση για να δούμε σε παγκόσμια επίπεδο, παγκόσμια οργάνωση υγείας και η ΦΑΟ ήδη. Το 2002 μας έχουν πει ότι για το πόσο υγιεινά και ασφαλή είναι τα προϊόντα Υποστηρίζουν λοιπόν αυτοί οι οργανισμοί ότι ο κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα ε, να χρησιμοποιεί ακίνδυνα τρόφιμα και γίνεται όμως στο τέλος και κάτι το επικειμενικό. Δεν είναι μόνο συλλογικό δικαίωμα. Είναι κάτι το οποίο ενισχύεται από το δικαίωμα ατομικά του καθένα να καταναλώνει τρόφιμα ακίνδυνα. Και βλέπουμε και την ομοθεσία την ευρωπαϊκή που έχει τεθεί υπέρ της προστασίας του καταναλωτή σε ένα επίπεδο πιο υψηλό και ισχύουν, έχουν επικρατήσει διάφορες ρυθμίσεις σε γενικό επίπεδο το οποίο όμως σε επίπεδο καμιά φορά διαστρεβλώνει την αγορά, στρεβλώνει την όλη αγορά και στο τελευταίο γύρο της Ουρουγουάης Έχουμε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για να υπάρξει μια κάποια ομοιομορφία και να έχουμε και τον πύχη σε τέτοιο ύψος που να ισχύει αυτό για όλες τις χώρες και παράλληλα με τα όσα ισχύουν στα διάφορα τρόφιμα και φυτοφαρμακευτικές επίσης ρυθμίσεις. Βλέπουμε λοιπόν την κάθε χώρα που έχει τα κατάλληλα όργανα που προσέχουν αυτό το επίπεδο αθότητος εισαγωγικά του τροφίμων, ακόμα και η Κίνα μπροστά στα διάφορα σκάνδολα διατροφής προσέχει αυτή την ε, ε, με ένα δικό της οργανισμό Food Drug Administration όπως τον Αμερικανικό προσέχει πια την κατανάλωση, τη διάθεση πρώτα και κατανάλωση μετά αυτών των τροφίμων. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο το διεθνές από το 1995 μέχρι τώρα είχαμε πολλές αντιπαραθέσεις ε, σε αυτά τα χρόνια, τα 15 τελευταία χρόνια. Και ανάμεσα στο 1995 και το 2001 είχαμε πάνω από 2.400 ε, υποθέσεις ε, με προβλήματα προϊόντων διατροφής οι Ρόμπερτς και Ανέβερ έκαναν ε, μία έρευνα που δείχνουν αυτές τις περιπτώσεις ε, και προσπαθούμε να τα βρούμε όλα αυτά σαν σημείο αναφόρας ε, για το τι γίνεται, ποια ήταν τα προϊόντα τα παθολογικά και τα τοξικά. Στο γενικό αυτό πλαίσιο Όπως είπε ο προηγούμενος εισηγητής, θα πρέπει να δούμε ότι έχει βυθιστοποιηθεί ιδιαίτερα για το πόσο γίνανε τα τρόφιμα. Έχει βυθιστοποιηθεί, επαναλαμβάνουμε, ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Και από το Ευρωμετρό στο τέλος Μαρτίου η κοινοτική κοινή γνώμη σαν πρώτη ανησυχία της στο γεωργικό τομέα έχει τα αθώα αυτό τρόφιμα, πως μπορεί να είναι ακίνδυνα, το 50% αυτό το θέμα προσέχει ανάμεσα στους καταναλωτές, του κοινωτικούς, στον αγροτικό, του γεωργικό τομέα. λοιπόν όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές περιπτώσεις ε, σχετικά με την ε, ασφάλεια των τροφίμων αντιμετωπίζει προβλήματα πολλές φορές ε, αντιπαραθέσεις, προσφυγές κλπ και προσπαθεί να λάβει μέτρα, γίνονται προσπάθειες ε, για μέτρα μη δασμολογικά, τα οποία όμως καταλήγουν σε προσπάθειες προστατευτισμού. Και αν ρίξουμε ματιά στα στοιχεία της Eurostat ανάμεσα στο 2000 και στο 2008, τι διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώπη είχαμε μια αύξηση κατά 43% των εξαγωγών, αλλά επίσης μια ιδιαίτερη αύξηση των εισαγωγών, άλλο τόσο περίπου σαν ποσοστό. Και έτσι έχουμε μια αφετηρία σκέψης για επανεξετάσουμε το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων και αυτό μάλιστα στα πλαίσια ευρύτερων διαπραγματεύσεων για τις πολυμερείς ε, συμφωνίες να δούμε και τι θέση μπορούμε να υποστηρίξουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αποτυχία και μετά των ε, διαπραγματεύσεων της Ντόχα για τα μέτρα, για τα τρόφιμα, από το 2006 μέχρι σήμερα όλες οι συναντήσεις που έγιναν εξέταζαν πάντα τις ε, ενισχύσεις ε, στις ε, εξαγωγές, τις εισαγωγές, τους δασμούς, όλα αυτά. Ενώ οι ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων δεν ήταν σημαντικό σημείο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της Ντόχα ο Επίτροπος Λαμή είχε επαναλάβει αρκετές φορές ότι θα ήθελε όλα αυτά να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2010 και το πολύ στις αρχές του 2011. Τώρα να δούμε τι γίνεται μετά από όλες τις διαπραγματεύσεις της Δημερής οι οποίες ε, διεξάγονται μετά από την αποτυχία του γύρω της Ντόχα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν μέχρι τις διαπραγματεύσεις του 2006 για το εξωτερικό εμπόριο δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στις διμερείς ε, διαπραγματεύσεις αλλά μετά το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει και πάλι σημασία ιδιαίτερη στις αυτές τις διμερείς διαπραγματεύσεις και το WTO, το, το WTO μας λέει ότι ο ΠΟΕ μας λέει ότι από τον ότι έχουμε αλλαγές, μάλλον έχουν ολοκληρωθεί 362 συμφωνίες εμπορικές και 211 ισχύουν ενεργά σήμερα. Όλες οι χώρες έχουν πολλές παρόμοιες κλήσεις συμφωνίες διμερείς εκτός από την Μογγολία από ό,τι ξέρω. Και αυτό τι μας δείχνει. Ότι όλα αυτά τα διαπραγματευτικά παίζονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα και θα πρέπει εκεί να ισχύσει η φιλοσοφία που διέπει την ε, ευρωπαϊκή γεωργία για την ασφάλεια τροφίμων, για την ποιότητα τροφίμων σε αυτά τα προϊόντα λοιπόν. Τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι οικονομολογοί. Τι θα γίνει ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των συναλλαγών ε, ε, πολύπλευρα και μονόπλευρα και πώς θα μπορούν να συνδυαστούν ε, αυτές οι δύο μέθοδοι και διαπραγματεύσεις. Πολλές ε, μελέτες δείχνουν ότι μακροπρόθεσμα σε διμερές επίπεδο συμφωνίες μπορούν να δημιουργήσουν ακριβώς δυσκολίες που μερικές φορές αναφέρονται σαν συμφωνίες μακαρονικές, ζυμαρικών και πέρα από αυτό που γίνεται για την ποιότητα που θέλουμε να προσφέρουμε σε διμερείς ή πολυμερείς συναντήσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε το παραγωγικό στυλ το ευρωπαϊκό και πώς αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να το φέρουμε στο Διεθνές Τραπέζι Διαπραγματεύσεων. Όλα αυτό το όλα αυτά τα ξέρουν όλα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και για τον σεβασμό στον κόντεξ αλιμεντάριο όπως είπαμε πριν από λίγο. Αλλά θα πρέπει να δούμε η παραγωγή Ευρωπαίοι τι ακριβώς θα πρέπει να σέβονται στην παραγωγή τους και όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής θα πρέπει όλα αυτά να τα σέβονται και οι τρίτες χώρες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά μας και θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το σύνολο κανόνων θα ισχύσει, επαναλαμβάνουμε, και για άλλες χώρες. Ε, αυτός ο διμερής χαρακτήρας, ο πολύπλοκος χαρακτήρας που θα ισχύσει για να προωθηθεί η ευρωπαϊκή αντίληψη επί του θέματος ε, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και στα δύο αυτά επίπεδα στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Ε, έτσι φαίνεται σαν κάτι το αυτονόητο, αλλά που δεν χρειάζεται κάτι να το επαναλαμβάνει. Ταυτόχρονα όμως να δούμε και την εξέλιξη του γύρου της Ντόχα. Χρειάζεται να δούμε να εξετάσουμε τις μελέτες και τις γνώμες των φορέων στον ΠΟΕ και να δούμε αυτόν ε, τον τομέα και ότι ο ΠΟΕ αναθεωρεί αυτήν την πολιτική της. Ποιος είναι ο στόχος. Οι δέσμοι μέτρων ε, για την ε, ασφάλεια των τροφίμων να είναι οι ρυθμίσεις όσο γίνεται πιο διάφανες και έχουμε διάφορα μέτωπα, όλο και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο και εκεί πιστεύουν αυτά τα μέτρα για τα τρόφιμα ε, και διάφορα μέτρα ακριβώς ε, άλλων χωρών αποτελούν ένα τρόπο παρεμπόδισης διεξαγωγής ελεύθερου εμπορίου. Ε, Εντάξει, κάτι που ίσως είναι λίγο προχωρημένο, αλλά το είδα και πολλές φορές να το λένε επιστήμονες και το άκουσα. Και είναι σαν κάποιος ψάχνει σε ένα φωτεινό δωμάτιο και πλησιάζει ένας αστυνομικός και του λέει «Μα τι έχασες» «Έχασα τα κλειδιά μου». «Ναι, αλλά πού τα έχασες τα κλειδιά σου» «Δεν ξέρω πού τα έχασα, αλλά εγώ τα ψάχνω εδώ». Εδώ ήταν το πιο φωτεινό μέρος και εδώ τα ψάχνω, επειδή είναι ευκολότερο να τα βρω αν τα έχω χάσει εδώ. Αυτό συμβαίνει. Πολλές χώρες ε, αυτό κάνουν. Αν εντάξει, ε, αυτά είναι τα μέτρα που απαιτούνται. Εδώ είναι που μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σχετικά με ε, ενισχύσεις, στήριξη κλπ. Ε, ενώ από την άλλη μεριά αυτά τα μέτρα είναι δύσκολο να ελεγχθούν παντού σε διάφορους χώρους, σε διάφορους τομείς αλλά εμεί τα ψάχνουμε σε ένα μόνο τομέα. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ήδη. Κάποιος θα μπορούσε να προτείνει αυτά τα μέτρα για τα τρόφιμα, για την ασφάλεια των τροφίμων, θα μπορούσε να προτείνει να μπουν σε μια κοινή δέσμη εξέτασης μέτρων μαζί με άλλες διαπραγματεύσεις για να δούμε τι συμβαίνει εδώ απέτυχε ο προηγούμενος γύρος της Ντόχα και τώρα καταβάλλονται προσπάθειες για περικοπές, το να το άλλο 48% έτσι με κατοστία ποσοστά. Ε, όλα αυτά για να συζητηθούν και πού θα τεθεί ο πύχης ε, από πλευράς της Ευρώπης για να θεωρεί ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή. Εδώ ακριβώς με ποιο τρόπο θα τα κάνουμε όλα αυτά λοιπόν. Ο δρόμος ποιος είναι. Να κινηθούμε σε μια διμερή λογική, εντάξει, δεν μπορούμε να απαλλαχθούμε από αυτήν. Και οι ίδιε οι Ηνωμένες έχουν αυξήσει αυτά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τις διμερείς συμφωνίες τους. Και στην Ασία, οι διάφορε ασιατικέ χώρε το έκαναν αυτό. περισσότερε διμερεί ε, συμφωνίες και θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν και την πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Αλλά όπως είπε προηγουμένως ο Επίτροπος, να δούμε πώς ε, την αξία μας θα την δείξουμε και θα την εφαρμόσουμε σε διμερείς Συναντήσει και διαπραγματεύσεις και σε τρίτες χώρες για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι τρίτες χώρες την αξία της δικής μας ε, πορείας και των δικών μας μέτρων. Μεσοπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα να μπορέσουμε να συγκλίνουμε με αυτές τις χώρες και να μπορέσουμε στη συνέχεια μέσω πολυμερών συμφωνιών να μπορέσουμε να τίνουμε περισσότερο προς μια προσέγγιση που να μοιάζει με την ευρωπαϊκή για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Το μεγάλο το πρόβλημα και η πρόκληση που θα ήθελα να σας πω εδώ είναι να καταλάβουμε εάν στις διαπραγματεύσεις της πολυμερής, στις μελλοντικές το θέμα της δέσμης αυτών των μέτρων, τι θα γίνει, θα υπάρξει μια ταυτόχρονη διαπραγμάτευση, ξεχωριστή διαπραγμάτευση σε σχέση με το σύνολο των διαπραγματεύσεων. Έχουμε επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι εάν πέρα από τους δεσμούς και με υψηλότερα πρότυπα, τι γίνεται, ποιος κερδίζει από αυτό, η παραγωγή, οι καταναλωτές, αλλά τελικά απαντήσεις ε, απόλυτα σίγουρες δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να δούμε πού πρέπει να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη δική μας την αντίληψη. Αυτή είναι μια πρόκληση που θα μπορούσε να είναι κάτι που θα μας κάνει να κερδίσουμε τη μάχη για το μέλλον το δικό μας της Ευρωπαϊκής ε, Γεωργίας και στο μέλλον. Ευχαριστούμε τη Μαριάντζελα Περίτο, λέει ο Πρόεδρος, την ευχαριστούμε για αυτήν την σημαντική εισήγηση και τώρα τελευταίος ε, εισηγητής εμπειρογνώμων είναι ο κύριος Αμπτελ Χακίμ Χαμουντή από το Ίνρατο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωπονικής Έρευνας που θα μας μιλήσει για τις διοικητικές σχέσεις ε, ανάμεσα στην κοινοτική ρύθμιση και τον γεωργικό τομέα. Αμέσως μετά τον κύριο Χαμούντι θα ξεκινήσει όλη η συζήτηση. Ήδη έχουν εγγραφεί συνάδελφοι να να βλάβουν το λόγο. Έχουμε αποδικατιστεί, μας έχει αποδεκατήσει μάλλον το σύννεφο της τέφρας από το ηφαίστειο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο κ. Χαμουντή έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αντέλ Χακίμ Χαμούντι, ονομάζομαι και εργάζομαι για το Εθνικό Ινστιτούτο Αγρό νομικής έρευνας. Και δεν θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα των διοικητικών περιορισμών των νομοθεσιών, των κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν στο θέμα αυτό και των περιορισμών ως προς την ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία, κοιτώντας το από την έποψη του μικροοικονομολόγου. Και θα προσπαθήσω να σας δώσω μια σειρά από υπόψεις για να δείτε κι εσείς ε, τις διαφορετικές πτυχές από τις, με τις οποίες, ε, από τις οποίες μπορεί να προσεγγίσει αυτό το ζήτημα. Ξεκινώ λοιπόν με το θέμα καταρχάς της νομιμότητας, νομιμοποίησης καλύτερα των κανονισμών που έχουν να κάνουν με την ε, ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων διατροφής. Σε τρεις πτυχές θα αντιχωρήσω σε μια διαδική προσέγγιση καταρχάς, εάν πρέπει να υπάρχει απαγόρευση ή όχι. Πρώτον, δεύτερον, εάν πρέπει, ποιο είναι το επίπεδο της προσέγγισης, το επίπεδο δηλαδή των προϋποθέσεων ή των απαιτήσεων εναντί του παραγωγού ή του καταναλωτού ή γενικά που ορίζει η κοινωνία. Και τρίτον, μέσα. απαιτησεων του παραγωγου η εργαλεία που αξιοποιούνται από τη στιγμή που η κοινωνία προσδιορίζει το επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων. Θα προσπαθήσω λοιπόν να εξηγήσω με πολύ σύντομο τρόπο την ε, νομιμότητα είτε ο θεμητών μια παρέμβασης με βάση κάποιες απαιτήσει τη κοινωνίας που δεν ε, απορρέει πάντοτε από την ίδια λογική ε, υπάρχουν οικονομικά πολλέ φορές κριτήρια κοινωνικές επιλογές μετά θα προσπαθήσω να προσδιορίζω την έννοια της ανταγωνιστικότητας με βάση δύο πτυχές του, του κόστους προσαρμογής στην νομοθεσία και το κόστος επί των αναμενωμένων εσόδων από τη στιγμή που θα έχει αναλάβει ο παραγωγός το ε, κόστος αυτό. Το κόστος προσαρμογής αυτό καθεαυτό δεν αρκεί για την αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου θα προσπαθήσω να εξηγήσω το πόσο διαγωνιστικότητα μπορούσε να ενισχυθεί και χάρη στην αναζήτηση μέσων που θα μειώνουν, ε, θα ελαχιστοποιούν το κόστος στην παραγωγή, αλλά και χάρη στην παρακολούθηση και συνεργασία με τους παραγωγούς και την ασθενή ε, παρακολούθηση και, και του ανταγωνισμού, έτσι ώστε το κόστος που εφίσταται ο παραγωγός να είναι αντίστοιχο και με την προσπάθειά του προσπάθεια την οποία καταβάλει για την ασφάλεια των τροφίμων. Για, την, ε, για το πόσο είναι θεμητό λοιπόν ε, να αναπτυχθεί μια δημόσια παρέμβαση, η απάντηση είναι ναι, απλούστατα γιατί είμαστε σε ένα πλαίσιο στο οποίο η αγορά δεν μπορεί αυτόματα να ρυθμίσει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας, επαρκές δηλαδή για την δημόσια υγεία. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν μπορεί η ασφάλεια των ε, διατροφικών αυτών γεωργικών ε, προϊόντων ε, να αρκέσει ως χαρακτηριστικό επαρκές ώστε ο καταναλωτής ε, να αρκέσει ω χαρακτηριστικό που θα επιτρέψει τον καταναλωτή να, διαλέξει ένα τέτοιο προϊόν, γιατί συνήθω δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την ασφάλεια ο καταναλωτή. Επίση, προσπάθεια για αξιολόγηση και ποσοτική αξιολόγηση τη αυστηρή ε, αρκετέ φορέ νομοθεσία και του κόστου που μπορεί να έχει αυτή, αλλά ταυτόχρονα και η αρχή τη πρόληψη την οποία έχει επιλέξει το κοινωνικό σύλλογο, ε, εξαρτάται από τη στάθμιση μεταξύ της ζήτησης, κοινωνική ζήτησης, της, επιστημονική επιστημονικής έρευνας, των δεδομένο δηλαδή της επιστημονικής έρευνας, η οποία βεβαίως θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα της κοινωνίας δεν θα προξενούν περιττό οικονομικά ή υπερβολικό κόστος. Θα είναι δηλαδή ευθυγραμμισμένα με την επιστημονική έρευνα, αλλά κατά βάση η επιλογή είναι επιλογή κοινωνική, του κοινωνικού συνόλου. Και άρα θα πρέπει όχι να μειωθούν οι απαιτήσει τη κοινωνία, εφόσον υπάρχει συνένεση φυσικά, αλλά να ε, προασπιστούμε και ενδεχομένω και να εξεγάγουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσει αυτές τη κοινωνία. Ω προ την επιλογή των μέσων ή εργαλείων. για την επιλογή τώρα των μέσων παρέμβαση, δημόσια παρέμβαση. Όταν προσδιοριστεί το επίπεδο ασφάλεια, το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλεια, η επιλογή των μέσων εργαλείων, η φύση του ή ο συνδυασμό αυτών μπορεί να προκαλέσουν και οικονομικό κόστο τόσο για τον νομοθέτη όσο και για τον παραγωγό. Φερρυπίν, καταμερισμός τη ευθύνη μεταξύ των διαφόρων τμήματων της παραγωγής, παραγωγής, η φύση των συστημάτων ελέγχου, οι ε, επιλογές σε σχέση με το αν θα είναι ε, εκούσια ή υποχρεωτική υπαγωγή σε κάποιους κανόνες δηλαδή κάθε είδους μέσο νομοθετικό, μέσο μάλλον ε, ή συνδυασμό μέσων μπορεί να έχει οικονομικό κόστος ή συνέπειες διαφορετικό ανάλογα και με την ασφάλεια που επιδιώκεται. Εξού και ο συνδυασμός αυτών των μέσων και εργαλείων είναι πάρα πολύ σημαντικός ως προς την ε, αποτελεσματικότητα της νομοθετικής ε, ή της κανονιστικής επέμβασης, παρέμβασης και βέβαια θα έχει διαφορετικό κόστος και για το δημόσιο αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα, παραγωγό και μη, αλλά και ως προς την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Αυτή την έπαψη λοιπόν. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις ε, παρουσιάσουν διαφορετικά μέσα, νομοθετικά αλλά όχι μόνο, που προσδορίσουν την ευθύνη των διαφορών παραγόντων και παραγωγών, αλλά και εθνικά μέσα που έχουν αυτό το χαρακτήρα της υποχρέωσης αποτελέσματος με βάση τα χαρακτηριστικά που επιδιώκονται προς το τελικό προϊόν. Δηλαδή επιτρέπει η ρύθμιση, επιτρέπουν οι ρυθμίσεις γενικά ένα ευρύ πεδίο διάκρισης διακριτικής ευχέρειας για τον παραγωγό με βάση την υποχρέωση αποτελέσματος. Αυτή η ελευθερία λοιπόν που επιτρέπεται στον ε, ιδιωτικό τομέα είναι λίγο πολύ η εκείνη η οποία ε, παρήγαγε αποτελέσματα και απαντήσεις τα οποία μετατράπηκαν με τη σειρά τους σε προδιαγραφές και ως προς τη μετατροπή, τα μεταποιημένα δηλαδή προϊόντα και ως προς την προμήθεια, τον καταναλωτή αλλά και τον προμηθευτή αυτών των προϊόντων. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι συλλογιστικέ, αλλά δεν θα επισέλθω σε αυτέ τι συλλογιστικέ των διαφόρων παραγόντων που είναι πολύ σημαντικέ βεβαίω προ την ε, παραγωγή των γεωργικών ε, διατροφικών προϊόντων. Υπάρχει η λογική της επισήμανσης λοιπόν των προϊόντων έτσι ώστε ο, ο, ο καταναλωτής να βλέπει την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή αλλιώς υπάρχει η λογική της ε, υποχρέωσης για τον παραγωγό ή τον μεταποιητή να τηρήσει μια σειρά από προδιαγραφές χωρίς αυτές απαραίτητα να είναι ορατές για τον καταναλωτή. Αυτά λοιπόν τα είδη επιλογών και κυρίως αυτές τις οποίες προέβησαν οι μεγάλες αλυσίδες των ε, ε, σούπερ μάρκετ οδήγησαν στην ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο των διαγραφών Global Gap και, τα, και άλλες οι οποίες οδήγησαν σε ευρύτατες εμβέλειες προδιαγραφές τόσο στην Ευρώπη αλλά και στη διάδοσή τους και βέβαια την ε, δυνατότητα επιλογής σε πρωτογενή γεωργικά προϊόντα που γνωρίζετε ότι είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει ο παραγωγός μέσα από αυτή τη νέα προσέγγιση για τα πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα αυτή τη στιγμή συνεπάρχουν ιδιωτικά πρότυπα, μαζί με τις δημόσιες παρεμβάσεις, ρυθμιστικές και άλλες και μάλιστα θεωρείται ότι είναι πολύ πιο δεσμευτικά από την ίδια την νομοθεσία. Μέσα λοιπόν από αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικών προδιαγραφών εντοπίζουμε το ζήτημα της, του κόστους προσαρμογής στην δημόσια νομοθεσία, στην, στο δημόσιο δίκαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κόστος προσαρμογής βεβαίως επηρεάζει και την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αυτών ομάδων διατάξεων. Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί το κόστος σε ποιο κομμάτι οφείλεται στη δημόσια παρέμβαση στις ιδιωτικές δεσμεύσεις. Και λόγω της ελευθερίας που επιτρέπει η νομοθεσία στον να αναπτύξει ο παραγωγός με, την, τον κώδικα καλής συμπεριφοράς ε, μιας επαγγελματικής ε, τάξεως που υποστηρίζουν οι ε, κρατικές αρχές ή με την υπαγωγή σε ιδιωτικού χαρακτήρα κανόνες συμπεριφοράς επηρεάζεται ιδιαίτερα και η πρόσβαση στις αγορές και γι' αυτό το λόγο και κατά τρόπο παράδοξο πρέπει να πούμε υπάρχει μάλλον περιορισμένη αξιολόγηση του άμεσου κόστους ως προς την ε, του άμεσου κόστους για την προσαρμογή στη δημόσια νομοθεσία πέραν κάποιων ενδεχομένων ε, μελετών που έχουν να κάνουν με την ε, αγορά HACCP. Δεν υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά μέθοδοι ανάλυσης ποσοτικές οι οποίες να επιτρέπουν να αξιολογήσουν πόσο κοστίζει άμεσα μάλιστα ε, απευθείας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι ιδιωτικού χαρακτήρα προδιαγραφές που επιβάλλονται στον παραγωγό. Απάξει λοιπόν και έγινε δεκτή η έννοια της αρχής της πρόληψης και τη ασφάλεια των ε, γεωργικών διατροφικών προϊόντων όπω έχει στο επίπεδο που έχει γίνει δεκτή, πρέπει να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστο προσαρμογή ευθυγράμμιση με τι προτεγραφέ αυτέ, το οποίο μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις αποκλεισμού ενό παραγωγού ή μείωση ανταγωνιστικότητα. Αποκλεισμό παραγωγού ε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Υπάρχει, έχει μελετηθεί με κάποιες δειγματοληπτικές μελέτες και επιτόπου έρευνες και είναι όλο και περισσότερο από απόρρια των ιδιωτικών προδιαγραφών επειδή ο ιδιωτικός και μικρός παραγωγός δεν μπορεί να ανθέξει το οικονομικό κόστος προσαρμογής σε αυτές τις προδιαγραφές. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες στρατηγικές αντιμετώπιση του κόστους. Καταρχάς υπάρχει η δυνατότητα να ενθαρρυνθεί ο παραγωγός ή η παραγωγή στην ανάπτυξη αυτών των κωδίκων καλή συμπεριφορά που όμως θα πρέπει να επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να προκαλούν επιπλέον επενδύσεις ή ε, δυσβάσταχτε επενδύσει. Δεύτερη λύση μπορεί, πρέπει να, αναζητηθούν μέσα τα οποία θα επιτρέψουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό κέρδος παραγωγικότητας ενσωματώνοντας στους κώδικα συμπεριφοράς και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά και τρόπο διαχείρισης μιας εκμετάλλευση, σε τη διαχείριση ποιότητα. Τρίτη πιθανή στρατηγική για την ελεγχιστοποίηση του κόστους ε, προσαρμογής ενίσχυση της ε, ενσωμάτωσης σε ομάδες παραγωγών και γενικότερα δραστηριοποίησης στις, ε, σε πρώιμες φάσεις της αλυσίδας και των ε, κωδίκων συμπεριφοράς που θα μπορούσαν και βέβαια αυθόρμητα να οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας αλλά και σε μείωση σε δεύτερη φάση της ε, του κόστους προσαρμογής στις προδιαγραφές. Αυτά ως προς το κόστος. Χρειάζεται λοιπόν μια προσπάθεια για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος. Ως προς την ανταγωνιστικότητα τώρα. Ανταγωνιστικότητα. Το να εξεταστεί μόνο από την άποψη του κόστους ε, το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να δώσει πλήρη εικόνα. Οι τομείς ε, χαρακτηρίζονται από ατέλειες αγορών με αποτέλεσμα ορισμένα προϊόντα η ασφάλεια ορισμένων προϊόντων είναι απολύτω συνδεδεμένη από το κόστο παραγωγή και οι αγορέ είναι όλο και λιγότερο ε, ενοποιημένες, όλο και περισσότερο κατακαιρματισμένες εκτός από κάποια προϊόντα. Και λόγω και της συγκέντρωσης, άλλωστε νομίζω το ε, ανέφεραν και οι προλαλήσαντες και συμφωνώ μαζί τους, λόγω λοιπόν της συγκέντρωσης στην ε, μεταποιητική και την εμπορική ε, το εμπορικό κυρίως στάδιο, με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και τις μεγάλες μονάδες μεταποίησης υπάρχει μεγάλη επίδραση από αυτή, αυτό το στάδιο στην ζήτηση και βέβαια και την ποιότητα των αγαθών και το κόστος του πρωτογενούς προϊόντος. Άρα υπάρχει μια μετακύληση σταδιακή, δειλή ίσως, από τον τύπο αγοράς που θα χαρακτηρίζαμε ως spot προς τους τύπους αγοράς ε, που χαρακτηρίζονται συμβατικοί τύποι, μεγάλης δηλαδή εμβέλειας. Και έτσι η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών συστημάτων ή της γεωργίας αφήνει τη θέση της ε, ε, σταδιακά στην έννοια της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων αλυσίδων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων. Δηλαδή, ο παραγωγός θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης, διάθεσης στην οποία θα συσσωμετωθεί. αν θα είναι εγχώρια ή διεθνής, εάν θα πρέπει να ε, υποταχθεί στις εσωτερικές μόνο ή και σε διεθνείς προδιαγραφές, εάν θα υπαχθεί στις ε, προδιαγραφές και τις απαιτήσει ενός μεγάλου ε, λιανοπολιτή. Όλα αυτά εξαρτάται. Ε, από όλα αυτά εξαρτάται η δυνατότητα, και η, ανταγωνιστικό, η δυνατότητα παραγωγής και η ανταγωνιστικότητα του παραγωγού. Δεν έχουμε εμπειρικές, επαρκή εμπειρικά δεδομένα έτσι ώστε να δούμε πώς μέσα σε κάθε ένα από αυτά τα κυκλώματα ε, παραγωγής μεταποίησης και ε, διάθεσης η λιανικής μπορεί να συμπεριφερθεί ή μπορεί να έχει ανταπόκριση ο παραγωγός. Τα πάντα βέβαια θα κρυθούν από τη δική του προσπάθεια και ως προς την ε, ασφάλεια των ε, γεωργικών προϊόντων διατροφής. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα ζήτημα και σε ένα βαθμό θέμει τον ανταγωνισμού, ενδεχομένω από χώρε οι οποίε δεν έχουν τι ίδιε προδιαγραφέ και απαιτήσει ε, ω προ την ασφάλεια των τροφίμων. Πέραν αυτού όμω, εγώ θα περιοριστώ στι ε, πιο χαρακτηριστικέ νομίζω περιπτώσει, δηλαδή τα λεγόμενα ανώνυμα προϊόντα, τα προϊόντα τα οποία ω ε, εκ τη ποιότητά του δεν παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι κάπω θα έλεγα ομοιογενή και δεν τα αναγνωρίζει σε σχέση με προϊόντα προερχόμενα από τρίτα κράτη ο καταναλωτής. Έτσι λοιπόν μπορεί να αποτελέσουν ε, εδώ κυκλώματα παραγωγή μεταποίησης, διάθεσης περί μεγαλύτερη ε, απειλή ω προ τον Ευρωπαίο παραγωγό. Και το, και υπογραμμίζω ότι αυτή η απειλή μπορεί να είναι θεωρητική. Θεωρητική διότι και πάλι με την υποτακτική έγκληση τα κυκλώματα αυτά στα οποία επικρατεί η μεγάλη, οι αλυσίδες λιανοπολιτών, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και προμηθευτών επιβάλλουν στον παραγωγό τι ε, τις προδιαγραφές, ιδιωτικέ προδιαγραφές ποιότητας που όμω ισχύουν και για τα προϊόντα που εισάγουν αυτές έξω από, την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από τρίτα κράτη δηλαδή με αποτέλεσμα ή μάλλον με στόχο η ποιότητα που καταγράφεται μέσα στην ε, αλυσίδα αυτή σούπερ μάρκετ ή χονδρικής προμήθειας να είναι ομοιόμορφη και έτσι τελικά ο προμηθευτής ε, έχει απόδοση αντίστοιχη με, αυτή των, αντίστοιχη με τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλει για την εξασφάλιση των, ε, της ποιότητας του προϊόντων του και γι' αυτό θα πρέπει οι ευρωπαϊκές αρχές να παραγνωρίσουν τη σημασία της λειτουργίας ανταγωνιστικότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των αγορών ως στοιχείο βελτίωσης της παραγωγικότητας. Τώρα, εάν δούμε τις ε, εισαγωγές που περνούν από από προμηθευτή, από εισαγωγέα δηλαδή, ο οποίο ε, δεν απαιτεί υψηλέ προδιαγραφέ ή ανιχνευσιμότητα, εχνηλασιμότητα σε σχέση με προϊόντα προερχόμενα από τρίτα κράτη. Εν προκειμένου, ο αθέμητο ανταγωνισμό, όπω αναφέρθηκε νωρίτερα, ναι, μπορεί να έχει σκληρέ επιπτώσει και λόγω αυτών των ε, των εισαγωγών και κυρίω σε σημεία ή σε περιοχέ Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν υπάρχει επαρκή έλεγχο κρατικό αυτών των εισαγωγών ή τη ποιότητά του. Έτσι λοιπόν για να αποφευχθεί η είσοδος τέτοιων προϊόντων που δεν έχουν ε, εξίσου αυστηρές προδιαγραφές για τον Ευρωπαίο παραγωγό χρειάζεται ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ομοιογενείς προδιαγραφές ε, για όλα τα προϊόντα που περνάνε τα σύνορά μας και αξιοπιστία εν γέννη του συστήματος. Άπαξ και ένα αξιόπιστο το σύστημα έχει διτό ρόλο και προστατεύει τον Ευρωπαίο καταναλωτή, τη δημόσια υγεία δηλαδή, και συγκεκριμενοποιεί το επίπεδο φιλοδοξιών του μοντέλου, των επιλογών δηλαδή της κοινωνίας ως προς το μοντέλο ασφάλειας των διατροφικών μας προϊόντων που απαιτούμε, που απαιτεί η Ευρώπη δηλαδή και ταυτόχρονα εξασφαλίζει και ένα σύστημα αξιόπιστο, αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και θεμητό ανταγωνισμό για τους ευρωπαίους παραγωγούς έναντι των αθέμητων εισαγωγών προϊόντων χαμηλής ποιότητας και ε, μηδαμινής ιχνηλασιμότητας. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν έχει επίσης να κάνει και με τη δυνατότητα εξαγωγής του ευρωπαίου παραγωγού ε, προϊόντων μη επώνυμων ε, προς χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει πολύ στι ποιοτικέ του απαιτήσει, δηλαδή είναι 10 χρόνια πίσω και ενδεχομένω αυτό μπορεί να αποτελέσει απειλή για τον Ευρωπαίο παραγωγό. Παράδοξο δε είναι το γεγονό ότι ακόμη δεν υπάρχουν αρκετέ ποσοτικές μελέτε οι οποίε να αποδεικνύουν το συσχετισμό απώλεια τμήματων αγορά σε τρίτε αγορέ και ε, αυστηρότητα των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων έστω και αν φαίνεται κάτι τέτοιο σχετικά προφανές εκ πρώτη όψεω. Για τέτοιου είδου αγορέ, λοιπόν, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε διαφορετικέ λύσει για την ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα των παραγωγών τη Ευρώπη. Η πρώτη θα πρέπει να μειωθεί το κόστος προσαρμογής, να βελτιωθεί η ε, παραγωγικότητα με ορθή κατάλληλη επιλογή μέσων. Η εμπλοκή των αρχών στις ε, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την εναρμόνιση των προδιαγραφών και την εξασφάλιση διόδων με ε, οδηγούς για τους κώδικες συμπεριφοράς, ιδιωτικούς και μη, ε, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε λίγο πολύ να κάνουν τα, οι, τα, οι μεγάλες αλυσίδες ως προς την επιλογή των προδιαγραφών, των μέσων εφαρμογής και τη στήριση των προδιαγραφών και τα αποτελέσματα τελικά που εξασφαλίσουν, νομίζω ότι θα μπορούσε να τα μιμηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεύτερον, η φύση των αξιοποιούμενων από την νομοθεσία μέσων έτσι ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα, είτε είναι αυτά εθελοντικά, είτε είναι δεσμευτικά, υποχρεωτικά, η ορθή δοσολογία μεταξύ εμπλοκής του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που και θα εξασφαλίζει καλή ποιότητα προϊόντα και θα επιτρέπει την πλήρη ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα και την ισότιμη κατανομή της αξίας σε κάθε κομμάτι αυτής της αλυσίδας παραγωγής ε, μεταποίησης και διάθεσης. Επίσης, ο στόχος της ε, υπεροχής στις ξένες αγορές, στις τρίτες αγοράς, ενός προϊόντος για το οποίο ενώ είναι ομοιογενές, δηλαδή δεν, είναι επώνυμο, μπορεί να ξεχωρίσει σε σχέση με τα ομοιογενή προϊόντα. Αυτό θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε περισσότερο, να το επιδιώξουμε, γιατί έτσι θα μπορούσε θα μπορούσαμε προσπάθειες που καταβάλει ο Ευρωπαίος παραγωγός να αναγνωρίζονται και από τον καταναλωτή. Και κλείνοντας αυτή την ομιλία θα ήθελα να πω ότι η επιλογή ποιότητα του ευρωπαϊκού, μάλλον η επιλογή του ευρωπαϊκού μοντέλου ποιότητα βεβαίω ε, αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό αίτημα, σε μια απέτηση της κοινωνίας. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα μοντέλο που πρέπει να προασπιστούμε με τα μέσα που χρειάζονται. Πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέσα, όπως έλεγα νωρίτερα, με ελαχιστοποίηση του κόστου για την κοινωνία, για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίως και για τις δημόσιες αρχές επίσης. Επίσης βέβαιον είναι πως το ευρωπαϊκό μοντέλο μπορεί ξεκάθαρα να αποτελέσει εγγύηση υψηλής ποιότητας, υψηλής διαφύλαξης της δημόσιας υγείας του καταναλωτή, εφόσον βεβαίως, όπως υπογράφηκε και νωρίτερα, υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις και ε, ιδιαίτερα ενισχυμένη έλεγχη των εισαγωγών, με τους ελέγχους στα σύνορα που αναφέρθηκαν και νωρίτερα. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και η τρίτη λύση, την οποία θα πρέπει να διερευνήσουμε, πιστεύω, είναι το κατά πόσον μπορούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα μακροπρόθεσμα και σε περίπτωση επανειλημμένων κρίσεων, αντίστοιχων με αυτές που είδαμε πρόσφατα, και αξία, παύλα, καταφύγιο για τις προμήθειες, για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα των παγκοσμίων αγορών. Εάν δηλαδή επαληθευτούν αυτές οι κρίσεις, η προσαρμογή, μάλλον ο Ευρωπαίος παραγωγός έχει ήδη τέτοια πρόοδο, ε, βρίσκεται σε τέτοια ακμή ως προς την παραγωγή και την ποιότητα της παραγωγής του, που μπορεί να έχει σε περίπτωση επαναλημμένων κρίσεων σημαντικό πλεονέκτημα ε, ως προς την προμήθεια προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Αμπτελχακή Μαχαμουντή. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να κάνουμε δρόμο για ένα σύστημα που θα ενημερώνει, θα πληροφορεί τους Ευρωπαίους πολίτες για τα στάνταρτ που χρησιμοποιούν και οι υπόλοιποι εκτός Ευρώπης. Τελειώσαμε με τους εισηγητές εμπειρογνώμονες και τώρα συζήτηση σε Κερέσκι, επειδή θα πρέπει να αναχωρήσει και μετά όλοι οι υπόλοιποι, Φερνάντες Γκαρσία, Ντανέλη κλπ. κλπ. Σε Κερέσκι. Ο κύριος Σεκέρσκι. Μιλήσαμε για τρεις τομείς, για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια των τροφίμων με τις υψηλές προδιαγραφές, αυτός είναι ο δεύτερος τομέας και ο τρίτος τομέας είναι το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο παραγωγής ε, προϊόντων διατροφής. Ε, το ισορροπημένο γεωργικό μοντέλο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τροφίμων. Έχουμε πολλές προκλήσεις και πολλές προσδοκίες. Κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι το πιο σπουδαίο από όλα αυτά. Ποιο έχει πρώτη στη σημασία. Το σημαντικότερο καταρχήν είναι η υλοποίηση των προδιαγραφών, ο σεβασμό των προδιαγραφών για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι άλλοι δύο τομεί. είναι δευτερεύουσε σημασία. Το πρώτο, ο πρώτος θα πρέπει να εφαρμοστεί, να έχουμε υψηλές απαιτήσει και να υποστηρίξουμε την υλοποίηση αυτών των υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Τώρα, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Ο Επίτροπος Τσόλος είπε ότι χρειάζεται καλύτερη θέληση. Δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε συγκεκριμένες απαιτήσει στους εταίρους μας. Και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να καλύψουμε και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Μπορεί όμως από μόνη της η αγορά να εξασφαλίσει την ασφάλεια αυτών των τροφίμων. Γιατί έχουμε και το θέμα των αξιών και πιστεύω ότι επειδή η αγορά ενδιαφέρεται κυρίως για την απόδοση, αυτές οι ψηλές προδιαγραφές θα πρέπει να επιβληθούν έξωθεν. Γιατί υπάρχει το θέμα της παρέμβασης εδώ, αλλά υπάρχει το θέμα των αποτελεσμάτων. Είπαμε ότι μερικές χώρες επιβάλλουν τα πρότυπά τους και προδιαγραφές τους στα κοινοτικά προϊόντα, αλλά Άλλε προδιαγραφέ και πρότυπα ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα. Και αυτό επιτείνει τη διαφορά μεταχείριση μεταξύ των κοινοτικών και των εξοκοινοτικών προϊόντων. Εμείς όταν θέλουμε να εξαγάγουμε τα προϊόντα μας δεν πρέπει να υποκείμεθα στις απαιτήσει των άλλων για να δεχτούν τις εξαγωγές μας. Εμείς γιατί να μην απαιτούμε κάτι αντίστοιχο από τους ε, εξοκοινοτικούς παραγωγούς. Αφού και εμείς όταν εξάγουμε το ίδιο κάνουμε. Πώς τώρα θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα κριτήρια. Φυσικά ε, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από την συνύπαρξη στην Ένωση γιατί η αξία μας και το βάρο μας είναι ενισχυμένο όλοι αποφασίζουμε, συναποφασίζουμε για τον προσδιορισμό αυτών των προδιαγραφών και μερικέ φορέ εμεί είχαμε προβλήματα εμπορικών συναλλαγών με τη Ρωσία, αλλά η βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύτιμη και σίγουρα το αποτέλεσμα καλύτερο από ό,τι αν δρούσαμε μόνοι μα. Έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα, πώ αυτέ οι ποιοτικέ προδιαγραφέ και αυτά τα υψηλά πρότυπα θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και για τα περιφερειακά, για τα τοπικά προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη αξία και που μερικές φορές δεν εντάσσονται στους, στα γενικότερα πρότυπα. Για τις τοπικές αγορές ισχύουν μερικές φορές διαφορετικοί κανόνες και η παραγωγή τέτοιων τοπικών προϊόντων μερικές φορές εξανίστανται και διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι τα γενικότερα πρότυπα επιβαρύνουν πολύ την παραγωγή τους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τους ε, παραγωγούς να ελευθερωποιήσουν το κόστος της παραγωγής, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και το θέμα των διανομέων, το θέμα της διαφύλαξης της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει με το στόχο της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς μας να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα. Υπάρχουν βέβαια τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, αφενός. Έχουμε αφετέρου όμως και κάποιες απειλές για το περιβάλλον από τη συγκέντρωση της παραγωγής. Τώρα, η συγκέντρωση της διανομής οδηγεί σε μονοπόλιο. Αλλά και το μονοπόλιο έχει αρνητικές συνέπειες στην αγορά. Και μάλιστα στην έκθεση Μποβέ αναφέρθηκε η προσπάθεια αποδυνάμωση αυτής της συγκέντρωσης και πάταξη των μονοπωλίων στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν προσεκτικά να τα κοιτάξουμε όλα αυτά γιατί δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε όλα. Το θέμα είναι σε τι θα δώσουμε προτεραιότητα εις βάρος κάποιου άλλου ίσως. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σιγκερέσκη. Γκαρσία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Υπουργό, την Ισπανίδα Γεωργίας, Προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Γεωργίας και τον Επίτροπο επίσης που είναι μαζί μας εδώ. Είναι μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι κάτι το σημαντικό γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε πάντα και τους δύο μαζί μπροστά σε αυτή την ομάδα εργασίας, την απόψινή. Να ευχαριστήσω επίσης και τους τρεις ε, εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι είπαν όλοι τους πράγματα ιδιαίτερα σημαντικά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί και μα ζητούν κάθε φορά που έρχονται εδώ ή που τους βλέπουμε εμείς ε, ότι θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό που τους ε, ε, επιβάλλουμε εμείς να τους επιτρέψει να ανταγωνιστούν όπως και όλοι οι υπόλοιποι σε άλλα μέρη. Γι' αυτό πληρώνουν τους φόρους τους και γι' αυτό μας εκλέγουν εμά σαν εκπροσώπους εδώ στο Κοινοβούλιο. Σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Επίτροπος ε, για τις διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ και τις διμερείς διαπραγματεύσεις. Ε, έχει δίκιο ο Επίτροπος που λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια εμπορικά και ότι είναι η απέτηση του ίδιου του καταναλωτή του Ευρωπαίου. Δεν καταλαβαίνω όμως εγώ πώς γίνεται τώρα εμείς να έχουμε ακόμα αυτό το εμπόδιο ότι τα κράτη-μέλη δεν προσπαθούν να γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες σε διμερές επίπεδο. Στην Ισπανία υπάρχει αντιπαράθεση μόνιμη στους παραγούς ε, τους Ευρωπαίους που ε, παραπονιούνται ότι οι Μαροκινοί παραγωγοί δεν το κάνουν. Ε, ο ένας λέει ότι είναι ε, ευθύνη των Ισπανών, αλλά εμεί έχουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα και στη θάλασσα και είναι πολύ λίγοι έλεγχη... Και γι' αυτό υπάρχει συνεχώς μια καταγγελία αυτών των παραβιάσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αν μπορούμε να έχουμε μια ομάδα που να ελέγχει τα σύνορα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα γίνει για να μπορέσουν να αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στα κράτη-μέλη. Είναι από αυτά που μας απασχολούν. Και ο τελευταίος που έλαβε το λόγο, ο κύριος Χαμουντή το είπε, ότι εδώ υπάρχει πραγματικά, παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Επίσης σε τρίτες χώρες ε, απαιτούμε όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει, είναι μια υποχρέωση από την άλλη μεριά για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, τους κοινοτικού παραγωγούς. Ε, με την κυρία Περόνη δεν συμφωνώ γιατί λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη η οποία θέλει να ικανοποιήσει τον καταναλωτή, τον κοινοτικό. Δεν ξέρω με όλες αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε εμείς ε, στην παραγωγή προϊόντων κλπ. τι κάνουμε. Αλλά δεν είναι ο στόχος μας ο καταναλωτής, γιατί ο Ευρωπαίος καταναλωτής, αν ήταν εκείνος ο στόχος μας, η παραγωγή τρίτων χωρών, ε, θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να σέβονται τα ίδια ακριβώς πράγματα για την διασφάλιση αυτή και την ποιότητα των τροφίμων. Θα πρέπει να έχουν ακριβώ τα ίδια που θα πρέπει να σέβονται ε, στα, για τα φαρμακευτικά και όλα τα παρόμοια. Δεν το κάνω όμω και μια χώρα όπως ε, το Μαρόκο, Όπω το Λονάτε, που χρησιμοποιείται σαν φυτοφάρμακο και όμω το χρησιμοποιεί και μετά εισάγει τα προϊόντα του. Εμεί το επιτρέπουμε με τις, με τις ε, συμφωνίε που έχουμε κλείσει μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται. Ουσιαστικά για το περιβάλλον επικίνδυνα προϊόντα προϊόντα, τους αφήνουμε να τα χρησιμοποιούν. Τι γίνεται, αλλά ο Ευρωπαίος καταναλωτής καταναλώνει. Τι κάνουμε και αυτό ζημιώνουμε τον κοινοτικό παραγωγό που δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα φυτοφάρμακα που ξέρω ότι μερικέ φορέ. Όπω ξέρετε ότι για τα σπεριδοειδή ακριβώ ε, το μιγάκι που τα καταστρέφει, ε, είναι εις των παραγωγών μα, α πούμε στην ε, Ιβυρική Χερσόνησο. Υπάρχει λοιπόν αυτό, προϊόν, αυτό το πρόβλημα. Ακούστε, ναι, ε, η γεωργία είναι στρατηγικός τομέας και επειδή υπάρχουν πολλοί που απασχολούνται εκεί για μια παραδοσιακή καλλιέργεια, την καλλιέργεια των ατάλων, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα σε λογική τιμή να παράγει για τον κοινωτικό πληθυσμό προϊόντα. Ακριβώς εδώ που λέει ότι θα πρέπει για την αλλαγή των τιμών, την αύξηση των τιμών να δώσουμε μάχη μας και θα πρέπει να δούμε και τα, ίσως τα μέσα, τα εργαλεία διαχείριση αγοράς που δεν τα έχουμε τώρα όμως δυστυχώ εδώ και πέντε χρόνια ε, Συνεχώ, σιγά σιγά βλέπουμε ότι τα καταστρέφουμε αυτά τα αποσύρουμε η προσθέμενη αξία και της κοινωτικής παραγωγής και της βιομηχανίας τροφίμων στην Ευρώπη είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία. Αυτά έχουν σημασία. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία. Εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και ο κτηνοτρόφος και ο παραγωγός και θα πρέπει ε, ταυτόχρονα και η αντίστοιχη βιομηχανία. Από τα σημαντικότερα πράγματα είναι να τους προστατεύσουμε αυτούς. Και όταν λέγαμε ακριβώς για αυτά τα λευκά κένα, εδώ λέμε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα της διανομής στον τομέα αυτό λοιπόν και στην παραγωγή την πρωτογενή θα πρέπει να το πούμε ανοιχτά, καθαρά. Να πούμε ότι αυτά που ισχύουν για τον ανταγωνισμό θα πρέπει να ισχύουν για όλου. Γιατί αν η φαρμακομηχανία έχει για τόσα χρόνια ε, μέχρι να γίνουν γενικά προϊόντα για όλου, αν μπορεί να προστατεύεται, γιατί γίνεται με την βιομηχανία των τροφίμων. Εδώ πολλέ μικρομεσαίε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει οι οποίε επενδύουν σε παρόμοιε προσπάθειε και μετά του ε, στείλουν στον τοίχο για τα προϊόντα αυτά στις αγορές. Αλλά αυτά γίνονται, εκεί γίνονται πολλές καταχρήσεις και ε, χάνουμε πολλές τις εργασίες στην Ευρώπη εξαιτίας αυτό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να το συλλογιστούμε και θα πρέπει να το συλλογιστούμε καλύτερα και εμείς αλλά και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε την κυρία Γκαρσία. Ο κύριος Δανέλης. Grazie, Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την σημερινή σας παρουσία, καθώς επίσης και τους εμπειρογνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε. Γίνεται όλο και πιο καθαρό ότι κάποιοι από τους βασικούς στόχους που έχουμε θέσει στην κοινή αγροτική πολιτική δεν συνοδεύονται από ανάλογη βούληση για στήριξη. Έχουμε επιλέξει για παράδειγμα ένα ποιοτικό και πολυλειτουργικό μοντέλο γεωργίας. Αυτό το μοντέλο για να δουλέψει σε μια ανοιχτή αγορά προϋποθέτει νομίζω δύο πράγματα. Πρώτο, ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταμείβει εν μέρη τον παραγωγό για το υψηλότερο κόστος παραγωγής, ιδίως προκειμένου για την παροχή δημόσιων αγαθών που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερο, προϋποθέτει ότι θα δίνεται η δυνατότητα στον παραγωγό να παρουσιάσει την ποιοτική διαφοροποίηση του προϊόντος του στον καταναλωτή με την απαιτούμενη γι' αυτό σήμανση. Και αυτό σήμερα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ετικέτα για την ευρωπαϊκή προέλευση του προϊόντος, διότι κάτι τέτοιο θα παρέπεμπε σε έμεση παρεμπόδιση του ελεύθερου εμπορίου. Ο παραγωγός δηλαδή στο σημερινό συνδυασμό ελεύθερης αγοράς, χαμηλού προϋπολογισμού για τη γεωργία και διεθνών εμπορικών υποχρεώσεων, μένει εκτεθειμένο σε συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Αυτή η έκθεση του παραγωγού διαφέρει ανάλογα με τον τομέα παραγωγής και το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να δίνει προτεραιότητα και στην προστασία του Ευρωπαίου καταναλωτή. Και πάλι όμως ο καταναλωτής δεν έχει στη διάθεσή του ένα τρόπο ενημέρωσης για την προέλευση ενός προϊόντος. Σε ό,τι δε αφορά τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, η υπάρχουσα πολιτική σήμανση οδηγεί περισσότερο σε παραπλάνηση του καταναλωτή παρά σε ενημέρωσή του. Διότι Πόσο γνωστό είναι στον καταναλωτή ότι η ετικέτα με την ένδειξη των γενετικά τροποποιημένων συστατικών δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση περιεκτικότητας μικρότερης του 0,9%, πόσο είναι γνωστό ότι δεν είναι καν υποχρεωτική όταν η παρουσία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών οφείλεται σε τεχνικά αναπόφευκτο γεγονός ή σε τυχαία επιμόλυνση και όλοι ξέρουμε ότι οι τυχαίες επιμολύνσεις είναι πολύ εύκολο να γίνουν και γι' αυτό άλλωστε είναι και τεράστια η απειλή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για τη βιοπικιλότητα. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ειλικρινεί ω προ την προστασία του καταναλωτή, επισημένοντα υποχρεωτικά μόνο τα προϊόντα που πιστοποιημένα δεν περιέχουν ή δεν έχουν επιμολυνθεί με γενετικά τροποποιημένου οργανισμού σε κανένα στάδιο τη αγροδιατροφική αλυσίδα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ποιε είναι οι πραγματικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή αγροτική πολιτική και την προστασία του καταναλωτή και πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλε αυτέ τι ανεπάρκειε αλλά και αντιφάσει, παίρνοντα υπόψη και βεβαίω του περιορισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Δανέλη Ζωζε Μποβέ και μετά Γκαρσία. Ναι, ευχαριστώ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, έφυγε βέβαια στο μεταξύ ο κύριος Επίτροπος. Νομίζω ότι άνοιξε η συζήτηση, άρχισε η συζήτηση, αλλά ξεχάσαμε στις διάφορες παρουσιάσεις και ομιλίες έναν σημαντικό παράγοντα που είναι η ενώση των καταναλωτών ή ενώσεις σωματεία αγροτών ή σωματεία προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί ποτέ το θέμα της ε, ε, υγειονομικής ποιότητας δεν θα είχαν τεθεί μόνο από τους ε, νομοθέτες αν δεν είχαν θέσει το ζήτημα κάποια κοινωνικά κινήματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις ορμόνες, μπορούμε να μιλήσουμε για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά κάθε φορά από έξω προέρχεται η αίτηση και η απέτηση για τη θέσπιση τέτοιων ρυθμίσεων. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχουμε πάρα πολλά θέματα επιτάπητος, δεν μπορούμε όλα να τα εξετάσουμε λεπτομεριακά. Για παράδειγμα το κρέας που είναι ε, καρπός ε, κλωνοποίησης, θα υπάρξει κοινοτική νομοθεσία σχετικά. Ήδη οι πολίτες αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτουν ε, τα προϊόντα που περιέχουν κλωνοποιημένο κρέας. Επίσης, το θέμα της χρήσης ε, νανοσωματιδίων στα τρόφιμα και αυτό το ζήτημα είναι ανοιχτό. Το γενετικό στροποποιημένο οργανισμοί επίσης αναφέρθηκαν. Και στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συζήτηση και ψηφοφορία για το ανασυντεθέμενο κρέας. Γιατί υπάρχουν μηχανισμοί για τη θρομβίνη που χρησιμοποιείται προκειμένου να ανασυνδεθεί αυτό το και τα προϊόντα αυτά που κυκλοφορούν σήμερα έχουμε νέα προβλήματα και μάλιστα έχουμε αυτά τα νέα προβλήματα για έναν πολύ προφανή λόγο. Στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών είτε στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου αλλά κυρίως στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου ο κώτεξ αλιμεντάριου δεν είναι πια ένας μηχανισμός που μας προστατεύει αλλά αντίθετα ένας μηχανισμός που διευρύνει τη δυνατότητα να κάνει κάτι που δεν υπάρχει στη γραφή υποχρεώσεων ποιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση του κόντες αλιμεντάριου, ε, προβλέπεται δυνατότητα χρήση 180 προσθετικών ουσιών στον ίνο. Ο κόντεξ αλιμεντάριου σήμερα δεν είναι πια κάτι δημοκρατικό, είναι το αντίθετο. Και οι εταιρείε, οι επιχειρήσει εκπροσωπούν τι χώρε στον κόντεξ Αλιμεντάριου. Και μάλιστα η Ελβετία, που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ω εκπρόσωπο στο κόντεξ Αλιμεντάριου εκπρόσωπο από τι ε, γεωργοχημικέ βιομηχανίε, από μεγάλε εταιρείε, από πολυεθνικέ. Αυτή είναι οι συμβαλόμενοι στο κόντεξ αλιμεντάριου. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν με τι προδιαγραφέ και με του κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είδαμε πολλέ φορέ και είναι μία από τις εξηγήσει των αποτυχιών που εντοπίσαμε και ακούσαμε και τις απογευματινές ομιλίες από διαπραγματεύσεις που δεν έχουν τελεσφορήσει μετά το γύρο της Δόχας και μερικές φορές ε, η γεωργία γίνεται ως ε, αντικείμενο συναλλαγής της παγκόσμιας συμφωνίας και πολλές φορές θυσιάζουμε την ευρωπαϊκή γεωργία στο βωμό άλλων δραστηριοτήτων που θα θέλαμε να περάσουμε στην αγορά. Και δυστυχώς εκεί υπάρχει πρόβλημα γιατί συστηματικά αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης έχουμε πολλά άλλα σημαντικά θέματα, γιατί έχουμε τους εισαγόμενους κανόνες, ε, κανόνες εισαγωγής. Γιατί είπα θέλησαν να μας εξαγάγουν ε, κρέας με ορμόνες. Επίσης όλοι γνωρίζουμε ότι το κρέας που εισάγουμε από την Αργεντινή και τη Βραζιλία έχει πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που το θίξαμε πολλές φορές και στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά και στις διμερείς συμφωνίες μπορούν να μας επιβάλλουν άλλους ε, νέους κανόνες που μας ευνηδιάζουν στη δική μας παραγωγή. Δεν το αναφέραμε βέβαια για το θέμα της ζάχαρης για παράδειγμα, γιατί στην Ευρώπη παράγουμε ζάχαρη. Εισάγουμε ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και εξαιτία ε, μια διεθνού συμφωνία είμαστε υποχρεωμένοι να εισαγάγουμε 20% τη ζάχαρη που χρειαζόμαστε και που καταναλώνουμε. Γιατί όμω στι διεθνεί συμφωνίε δίνουμε δικαιώματα εξαγωγή ε, ε, ζαχάριος σε χώρες που δεν είναι παραγωγές, παραγωγή, για παράδειγμα στο Πέρου, τέτοιε συμφωνίε είναι κατάλληλε. Και για να γίνει μια παρισορρόπηση είναι και ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό. Αν μιλούμε για τι δικέ μα ρυθμίσει και του κανόνε, θα πρέπει να βρούμε το σωστό όριο και τη σωστή ισορροπία. Και χρειάστηκε με ενίσχυση, αλλά θα πρέπει και ο οικονομικό τελεστή Ευρώπη να παίξει το παιχνίδι όταν εξάγει. Για παράδειγμα, τα κατεψυγμένα πουλερικά που επιδοτούνται για πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από μία επιχείρηση όπως η Γαλλική Ντου που εξάγει στην Αφρική. Από όλες τις μελέτες που έγιναν για τις αφρικανικές αγορές φάνηκε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί για την κατάψυξη, τη σωστή κατάψυξη αυτού του κατεψυγμένου κρέατος, οπότε το προϊόν φθήρεται πολύ γρήγορα. Βέβαια, τέτοια πουλερικά εμείς δεν τα καταναλώνουμε γιατί τα πουλερικά αυτά τα μεγαλώνουμε σε τρεις εβδομάδες. Είναι ουσιαστικά προϊόντα που παράγονται μόνο για εξαγωγή προ τρίτε χώρε, προ φτωχέ χώρε, αναπτυσσόμενες χώρε. Εμεί τα θεωρούμε ακατάλληλα. Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να εξάγουν προϊόντα που εμεί τα κρίνουμε ακατάλληλα προ κατανάλωση. Νομίζω ότι δεν είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Είμαι υπέρ των αυστηρών κανόνων, αλλά να τις δέχονται όλοι και να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όταν είναι αυστηροί και για τις εισαγωγές και για τις εξαγωγές. Ευχαριστούμε τόσο, Μποβέ. Γκρασία Περές. Ευχαριστώ. Ε, Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρωτοβουλία διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου και να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Επιτροπής, ε, την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τους εμπειρογνώμονές μας και να πω ότι πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, μια κρίσιμη στιγμή που επιτέλους ε, αρχίζουμε μια συζήτηση με συγκεκριμένες προτάσεις επιτάπητος. Γιατί αυτή η πραγματικότητα δεν είναι καινούρια, την είχαμε αναφέρει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά Πιστεύω ότι σήμερα με τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου, με τη δράση της Ισπανικής Προεδρίας και με τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καταφέρουμε επιτέλους να δώσουμε μία απάντηση σε πολλούς άγνωστους χι και πολλά προβλήματα που έχουμε θίξει. Είμαι βέβαιη ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι πλεονέκτημα αυτή η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Είναι πολύ θετικές αυτές οι προδιαγραφές ποιότητας των προϊόντων, ευημερία των ζώων, σεβασμού του περιβάλλοντος. Σίγουρα είναι θετικά όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι αυτές οι αυστηρές προδιαγραφές ε, οδήγησαν σε μια απώλεια τη ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων γεωργών και κτηνοτρόφων. Αυτό το γνωρίζουμε, γιατί αυτό μας διαβιβάζουν σε κάθε ευκαιρία οι συμπολίτε μας γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Είναι σημαντικό λοιπόν στη συζήτηση αυτή για το μέλλον της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής να πούμε ότι σήμερα περισσότερο από, ποτέ και εξαιτία αυτή τη πραγματικότητα δικαιολογείται μια ισχυρή κοινή γεωρική πολιτική, μια όμω κοινή γεωρική πολιτική που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στι νέε προκλήσει και στη νέα πραγματικότητα. Υπάρχει τεράστια βεβαιότητα και θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε τον κλάδο. Γιατί είπαμε ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία έχουν στρατηγική σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα και να λάβουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Έχουμε επίγνωση ότι οι Ευρωπαίοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι προσφέρουν ένα κοινό αγαθό και για αυτή τους την προσφορά θα πρέπει να ανταμυφθούν. Γι' αυτό και δικαιολογείται περισσότερο από ποτέ η κοινή γεωργική πολιτική. Επίσης θα πρέπει να εξηγήσουμε και στους Ευρωπαίους πολίτες πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές ότι θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις και να εξεταστούν τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνηση, της ε, επέκτασης των ε, ποιοτικών προδιαγραφών και τη συμπερίληψή τους στις εμπορικές συμφωνίες. Επίσης, προαγωγή και διαφήμιση των ε, κοινοτικών προϊόντων, στήριξη των ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης ενίσχυση της ε, οικονομικής βιωσιμότητας της γεωργίας, αναζήτηση της ισορροπίας χωρίς ε, έγερση εμπόδιων και φραγμών. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει όχι μόνο να καταφέρουμε να τα αποτυπώσουμε σε ένα χαρτί, να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά να βρούμε τρόπους για να τους δώσουμε σάρκα και ωστά και να εφαρμόσουμε και στην πράξη όλες αυτές τις προτάσεις. Και ελπίζω ότι στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργό Γεωργίας θα συγκεντρωθούν όλες οι δυνάμεις ε, και δεν θα αφιστούμε προσπαθειών προκειμένου να αναζητήσουμε τις λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και όπως είπα υπάρχει τεράστια βεβαιότητα στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της Ένωσης. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν ένα μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους δώσει αμέριστη υποστήριξη και αναγνώριση για το, την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και για τις ποιοτικές προδιαγραφές. Θα τους υποστηρίξει όμως ταυτόχρονα ώστε η απώλεια ανταγωνιστικότητας να μην δημιουργήσει και στο μέλλον προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Καρσία Περέζ. Ναι, από κοινού εργαζόμεθα με το Συμβούλιο για την παρότριση αυτή. Όσλιν και μετά Μαγκίνες. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, είναι κάπως διχασμένη η συζήτηση ως προς την ε, ορθολογική της. Δηλαδή άλλοι ζητούν, ε, αφενός μεν ζητούμε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου όπως και ξεκάθαρα ο Επίτροπος αποδεικνύεται ότι ε, οι υψηλέ προδιαγραφές αποτελούν λόγο απώλειας αγορών. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τελικά τι θέλουμε. Οι υψηλές προδιαγραφές είναι ασφαλώς εγγύηση για τον ε, καταναλωτή μας και διατήρηση και τρόπος διατηρήσης της παραγωγής εδώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσαμε για τις παγκόσμιες αγορές. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε και σαφές ότι το 90% των παραγωγών μας δεν έχουν σχέση με τις παγκόσμιες αγορές, διεθνείς αγορές δεν βγάζουν τα προϊόντα του στο εξωτερικό και στι τρίτε χώρε. Άρα λοιπόν θα πρέπει νομίζω να δώσουμε την προσοχή μα ακριβώ εκεί που χρειάζεται, εκεί ακριβώ που είναι και τα συμφέροντα τη πλειονότητα των Ευρωπαίων ε, γεωργών και παραγωγών. Επίσης είδαμε από πολλές από τις ομιλίες που ακούστηκαν σήμερα ότι είναι ένα ύψιστον προδιαγραφών μοντέλο το ευρωπαϊκό μοντέλο. Υπάρχουν πολλά θέματα βεβαίως τα οποία θα πρέπει να διατυπωθούν επικρίσεις προς το ευρωπαϊκό πρότυπο παραγωγής. Έχουμε μαζικές συγκεντρώσεις ως προς την εκτροφή των ζώων που δεν εξυπηρετούν βέβαια τους όρους της ε, ευημερία ή της προστασίας των ζώων. Είναι πολλοί οι κανόνες που θα πρέπει να αλλάξουν αλλά γενικά νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε καλές ε, εξελίξει. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να δώσουμε την έμφαση και την εστίαση του ενδιαφέροντό μας στον παραγωγό, εκείνον ο οποίος έχει χάσει και από, την, ε, και από το εισόδημά τα τελευταία χρόνια και αυτό πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο του ε, ενδιαφέροντός μας. Για τις διεθνεί συμφωνίες. Νομίζω ότι η ραγδαία αύξηση των διμερών συμφωνιών ε, σημαίνει τελικά αποδιάρθρωση των προδιαγραφών για τη γεωργία. Εξυπηρετούνται δηλαδή ορισμένα συμφέροντα και όχι οι προδιαγραφές του γεωργικού τομέα. Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω κάτι για την ε, κυρία Υπουργό, διότι τίθεται το ερώτημα εάν τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ιδιαίτερω προξενούν πολλές ανησυχίες στην Ισπανία. Έχουμε πολλές ε, καταγγελίες για ανεπαρκή σήμανση προϊόντων που έχουν ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή έχουν, ε, στους οποίους έχουν συμβάλει γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί οι περιοχές όπου καλλιεργούνται αυτοί δεν έχει δώσει η ισπανική κυβέρνηση ικανοποιητικέ ε, απαντήσεις. Πολλές φορές έχουμε απευθύνει ερωτήσεις στην κυβέρνησή σας αλλά δεν έχουμε λάβει. Ελπίζω να μπορέσετε να το πράξετε εσείς σήμερα Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, ως κύριο χαρακτηριστικό ότι πρέπει να έχουν μια θέση στον ήλιο όλοι και όχι μόνο αυτοί οι οποίοι επιλέγουν το μοντέλο των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ευχαριστούμε οσλίν ε, Μαγκίνες τώρα. Η κυρία Μαγκίνες λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και το Συμβούλιο και την Επιτροπή και βέβαια όλους τους εδώ παρόντους και ομιλητές. Θα ήθελα ξεκινώντα να θέσω ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένω έθιξαν και κάποιοι άλλοι και μέσω, αλλά με αφορά ιδιαίτερω και άμεσα, ω προ μια απόφαση που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επανειακίνηση μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τι χώρε Μερκασούρ. Και παρά τι ίδιε τι ε, προειδοποιήσεις προς την Επιτροπή ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και θα οδηγήσει σε ε, σημαντικά προβλήματα το χώρο της γεωργίας και της κτηνοτροπηθίας, βλέπω ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση ούτε σε επίπεδο καν κοινοβουλίου για τα προβλήματα που θα προξενήσει αυτή η συμφωνία. Παρακαλώ λοιπόν και την Επιτροπή και το Συμβούλιο ιδιαίτερα η έμφαση και προσοχή να δώσουν στις επιπτώσεις που μπορεί αυτή η συμφωνία να φέρει για διάφορους τομείς της ε, παραγωγής μας, της γεωργικής, κτηνοτροφικής και τα μέτρα βεβαίως θα πρέπει να προβλεφθούν για τη στήριξη των παραγωγών μας. Οι προδιαγραφές επίσης θα ήθελα να επισημάνω δεν είναι μόνο ασφάλεια τροφίμων και επικεντρωνόμενη στην ασφάλεια των τροφίμων. Ε, χάνουμε μεγάλο κομμάτι της ιδέας των προδιαγραφών που είναι η βασική μας ασφάλεια. Ε, έχουμε πολύ σοβαρά μελήματα να ε, καλύψουμε πριν επικεντρωθούμε μόνο στην ασφάλεια των τροφίμων. Ειδικότερα δε όσον αφορά τις διμερείς εμπορικές ε, συμφωνίες δεν είμαι καθόλου πεπισμένη ότι πρόκειται να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε τι υψηλέ ευρωπαϊκέ μα προδιαγραφέ ε, στο μέγιστο. Είδαμε από το παρελθόν ότι υπάρχουν πολύ κακέ επιδόσεις. Για το Μαρόκο και τα ζυζανιοκτώνα έκανε λόγο η συνάδελφο, υπάρχει ζήτημα και με την Αργεντινή και με το Βόλιο κρέα. με δεκάδε χιλιάδε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ερωτήσει που έχουν πεθύνει στο Συμβούλιο και που αποδεικνύουν ότι, έχουν μειώ... Ε, ότι έχουμε μειώσει με την, ε, υπαγω... με την υποτίμηση των προδιαγραφών μα, τον αριθμό των εκμεταλλεύσεών μας στις χίλιες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα είδος αρχαίας τραγωδίας. Έχουμε όλοι τι ψηλές προδιαγραφές, όλοι ισχυριζόμαστε ότι θα τη στηρίσουμε και οι κυβερνήσεις και όλοι, αλλά η τραγική ηρωνία είναι ότι δεν προστατεύουμε τον παραγωγό μας εναντί των εισαγωγών, οι οποίες δεν είναι υποχρεωμένες να τηρήσουν τις ε, ε, προδιαγραφές αυτές και βέβαια η αγορά δεν είναι διατεθειμένη να καταβάλει το σχετικό τίμημα για τα ζυζανιοκτώνα και χαίρομαι ιδιαίτερω για τη σχετική απόφαση που λήφθη. Έκανε πολύ καλή δουλειά το Κοινοβούλιο. Εάν όμως επιτρέψουμε την παραγωγή ε, από τρίτες χώρες ή ε, χρήση ουσιών που είναι απαγορευμένε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι έχουμε λύσει κανένα πρόβλημα. Και πρέπει ιδιαίτερα να μα απασχολήσει αυτό. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την εφημερία των ζώων, και άκουσα και τι παρεμβάσει για υψηλέ προδιαγραφέ εφημερία ζώων και μελήματα. Και εμεί βεβαίω οι βουλευτέ ιδιαίτερα μα ενδιαφέρουν αυτό. Αλλά η παραγωγή αυγών σε κλοβού ω σύστημα πρόκειται υποτίθεται να καταργηθεί ε, σύντομα. Αλλά δεν ξέρω αν τα κράτη-μέλη έχουν λάβει τη σχετική, τη σχετική, μέρημνα για να θέσουν εφαρμογή την απαγόρευση. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι από ό,τι μα λένε ότι θα εξαχθούν οι κλοβοί σε τρίτες χώρες και θα εισαχθούν προϊόντα αυγών. Γιατί είναι τόσο υψηλό το κόστος για το καλύτερο, για τους καλύτερους τρόπους ε, οι πιο περιβαλλοντικούς οι πιο σωστούς τρόπους παραγωγής αυγού που δεν μπορούν να ανθέξουν τη μετατροπή στη νέα, στις νέες αυτές συνθήκες παραγωγής. Το ίδιο και για το χείριο κρέας και για πολλά άλλα. Αυτό είναι το πρόβλημα της ε, ασυνέπειας που έχουμε στην Ευρώπη. Ότι θέλουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, έχουμε υψηλέου στόχους και προδιαγραφές, αλλά το κόστος είναι τεράστιο για τον παραγωγό και τελικά καταλήγουμε, εάν δεν προσπιζόμαστε τις προδιαγραφές και τα συμφέροντα των παραγωγών μας, να εισάγουμε μόνο χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα. Και δεν ξέρω ποιο το είπε νωρίτερα. Το θέμα είναι νομίζω η επιλογή. Η κοινωνία μα ναι έχει επιλογέ αλλά πρέπει να είναι διτεθειμένη να κατεβάλει και το σχετικό τίμημα και σε αυτό νομίζω θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο εντό εισαγωγικών επιθετικοί, δηλαδή πιο σαφεί και απερίφραστη ενάντια του καταναλωτή όταν του μιλούμε για τι προδιαγραφέ. Τι ζητάει ο καταναλωτή, τι ζητάει η λιανική πώληση, τι ζητάει ο παραγωγό και ποιο τελικά πληρώνει. Αυτή η συζήτηση ασφαλώ θα πρέπει να γίνει. Τώρα σχεδιάζουμε το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική. Η... Όλη η συζήτηση νομίζω θα έχει να κάνει με την διασύνδεση των πληρωμών στο μέλλον με περισσότερο με τι περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ και γενικά υψηλότερε προδιαγραφέ ποιότητα. Αλλά αυτό σημαίνει και κόστο προσαρμογή για, τον... για τον παραγωγό και ενδεχομένω χαμηλότερη παραγωγή. Χαμηλότερη ποσότητα παραγωγή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε. Και όταν μιλούμε για ασφάλεια τροφίμων εδώ στο Κοινοβούλιο, πρέπει να βλέπουμε ταυτόχρονα και τη διάσταση της επαρκούς προμήθειας σε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύο, δύο οι διαστάσεις του προβλήματος και δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη μία ισόφελος της άλλης. Ξέρω, Πρόεδρε, ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι ένα ζήτημα όμως ζωτικό για τους παραγωγούς μας. Η ιδέα δηλαδή να έχουμε ύψιστες προδιαγραφές ποιότητας, τις οποίες θα τηρούν οι ίδιοι τις οποίες οφείλουν να πληρούν οι ίδιοι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να τους πείσουμε ότι δεν θα εισάγονται προϊόντα με, ε, που έχουν παραχθεί με πολύ διαφορετικό επίπεδο προδιαγραφών, με πολύ διαφορετικές συνθήκες. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το άκουσα και από τους ομιλητές σήμερα, το έχουμε δει και άλλες φορές. Δεν μπορούμε ως προς την ασφάλεια της ποιότητας των τροφίμων μας να κάνουμε συμβιβασμούς δεν χωρεί συμβασμό στο θέμα αυτό. Βεβαίω έχουμε την ηλεκτρονική σήμανση και τα ενότια και πολλά άλλα συστήματα που ίσω δεν εξασφαλίζουν την απόλυτη ασφάλεια τροφίμων, αλλά τελικά κοστίζουν και κάποιο πρέπει να υποστεί το σχετικό τίμα, να καταβάλει το κόστο αυτή τη ποιότητα. Ανησυχώ λοιπόν ιδιαίτερω γιατί μίλησα και για τι διμερεί δυνατότητε, διμερεί εμπορικέ συναλλαγέ, συμφωνίε καλύτερα. Συμφωνώ με τον κύριο Διαφωνώ γενικά με τον κύριο Μποβέ, αλλά σήμερα μπορώ να πω με χαρά ότι συμφωνώ ότι ε, το τίμημα θα είναι, θα το επιφορτιστεί η ίδια η Γεωργία. Ευχαριστούμε τη Μαγκίνες. Τελευταίοι δύο μιλητές τώρα. Γιάρ και Γκαβρόσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την ανταγωνιστικότητα της ε, παραγωγής τροφίμων, γεωργικής παραγωγής τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ορισμένοι δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν καλύτερα να δουν τα πράγματα σε όλες τους τις διαστάσεις. Έχουμε λοιπόν την ε, ε, διάθεση των προϊόντων την οποία αναλαμβάνει η αγορά, η οικονομία, αλλά τις προδιαγραφές τις ορίζουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε εν τέλει και τη σχετική ευθύνη και πολλοί διαπιστώνουν ότι οι προδιαγραφές πρότυπα δεν είναι θείοι νόμοι, είναι όροι τους οποίους ορίζουν οι πολιτικοί με κάποιο τρόπο. Αυτό πρέπει να το δούμε λοιπόν, αυτό το πλαίσιο, αυτά τα δεδομένα και να αντιληφθούμε ότι όταν βάζουμε ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι, για να είναι πιο φτηνό πρέπει κάπου κάποιος να έχει παραβιάσει συνθήκες ανταγωνισμού ή θεμητού ανταγωνισμού. Και ναι, έχουμε την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική παγκοσμιοποίηση, οικονομική παγκόσμια διαδικτύωση, αλλά ταυτόχρονα ο γεωργός δεν μπορεί να είναι ε, συνδεδεμένος ε, με κάποιον άλλο παγκόσμιο γεωργό ή παγκόσμια γεωργία. Πρέπει να δούμε όμως ότι όταν παράγεται σε μια περιοχή κάτι επηρεάζει αντίστοιχα η ποιότητά του, η έλλειψη ποιότητάς του και τα προϊόντα και την παραγωγή σε κάποια άλλη περιοχή. Όταν έχουμε λοιπόν απαγορευμένα προϊόντα μέσα σε ένα είδος μου τροφής, θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν υπάρχουν ή όχι. Ναι, αλλά δεν αρκεί το να έχουμε μια ετικέτα που θα μας λέει ε, υπάρχουν ε, επικίνδυνες ουσίες μέσα ή όχι. Γιατί ναι, όταν, ε, πάρω, όταν πάω να αγοράσω από τον Ευρωπαίο παραγωγό μία φράουλα, ένα, ένα κιλό φράουλες, μπορεί να μην υπάρχουν τα απαγορευμένα ζανιοκτώμα μέσα αυτές, αλλά όποιο θέλει να αξιοποιήσει τις φράουλες με τα απαγορευμένα ζανιοκτώμα θα βρει άλλε διεξόδους. Αυτό είναι βέβαιο. Και άρα θέλουμε όχι μόνο υγιή καθαρά τρόφιμα αλλά και συνθήκες ε, βιώσιμης σωστής παραγωγής όπως και για την κτηνοτροφία συνθήκες ευημερίας των ζώων. Επίσης, όταν προσδιορίζονται προδιαγραφές ή κίνητρα ενδεχομένω για την κοινή γεωργική πολιτική, δεν αρκεί αυτά να επιβάλλονται μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι της δουλειάς τελευταία ανάλυση, γιατί υπάρχουν οι μηχανισμοί του ελέγχου και της επιβολής των διατάξεων. Αλλά πρέπει οι απαιτήσει οι οποίες προσδιορίζουμε για τη δική μας εσωτερική αγορά, για το δικό μας εσωτερικό παραγωγό, να ισχύουν και προς τα έξω. Και εδώ χρειάζεται περισσότερο να κάνουμε προσπάθεια έτσι ώστε να ε, αντιμετωπίσουμε τις πολλές δυστυχώς παρεκκλήσεις και τις πολλές επίσης αδικίες. Και παραλαμβάνω, πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ διατάξεων, ρυθμίσεων δηλαδή και ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστούμε. Τελευταίος, μετά η Υπουργός κυρία Σπινόζα θα έχει το λόγο. Έχετε το λόγο εσείς. Ο κύριος Γκαβρόνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα όλοι ως την Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούμαστε με τη γεωργία και οι πολίτες μας που γνωρίζουν τη γεωργία ξέρουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και ξέρουμε ότι ισχύουν πολύ αυστηροί κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων, για το περιβάλλον και όλα αυτά είναι πολύ θετικά για τη γεωργία. Παρ' όλα αυτά, πολλά θα πρέπει να κάνουμε στον τομέα της γεωργίας και εντός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αλλά κυρίως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο που και η κυρία Υπουργό και ο κύριος Επίτροπος μίλησαν για την ανάγκη επέκτασης ε, διεύρυνσης και εξαγωγής και των ποιοτικών μας προδιαγραφών προς τα έξω και της ε, επέκτασης του γεωργικού ευρωπαϊκού μοντέλου και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δυστυχώς πολύ θα περιμένουμε μέχρι να εφαρμοστούν αποτελεσματικά όλοι αυτοί οι κανόνες ε, και παγκοσμίω. Και στο μεταξύ μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ε, πολλοί από τους παραγωγούς μας και να σταματήσουν πια να παράγουν. Αναφέρθηκε πολλές φορές ε, η ανάγκη για αποτελεσματικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των κανόνων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερες προσπάθειες, δηλαδή στην εφαρμογή και στην εκτέλεση. Υπάρχει όμως ένας τομέας στον οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Είναι ένας ε, τομέας που είναι σημαντικός για ολόκληρη την γεωρική παραγωγή. Γιατί πολύ πιθανόν να χάσει την ανταγωνιστικότητά της η γεωργική παραγωγή και όχι εξαιτία των κανόνων. Στην Ουκρανία, μετά τις εκλογές, έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά της πολιτικής, αλλά ε, δεν έχουν γίνει καθόλου αλλαγές και σε ό,τι αφορά την οικονομική σύνδεση της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να θέσω την ερώτηση προς τον Επίτροπο βέβαια, αλλά τι θα γίνει, η Ουκρανική Γεωργία θα ενταχθεί στην ε, κοινή αγορά. Γιατί η Ουκρανία έχει σημαντική γεωργική παραγωγή και μάλιστα παραγωγή Είναι πολύ μεγάλη σιτοπαραγωγός χώρα και αν ενταχθεί η Ουκρανία στην ε, ενιαία αγορά δεν υπάρχει περίπτωση να ανταγωνιστεί την Ουκρανική παραγωγή ούτε η Γαλλική ούτε η Γερμανική. Και μάλιστα μαζί με τη Ρωσία φέτος η Ουκρανία θα παράγει 50 εκατομμύρια τόνους ε, σίτου Αποκλείται να αντισταθούμε στον ουκρανικό ανταγωνισμό αν συνδεθεί με την ενιαία αγορά η ουκρανική οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια πολύ διεξοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα έχει μια τέτοια απόφαση στην κοινοτική γεωργία, εφόσον φυσικά υιοθετηθεί μια τέτοια απόφαση. Σήμερα αναφέρθηκε το θέμα της ενημέρωσης προς τους καταναλωτές, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε και την πληροφόρηση προς τους παραγωγούς μας. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα για τους ε, γεωργίους της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύνδεση της ουκρανικής οικονομίας στην ενιαία αγορά. Θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Δεν μπορεί να γίνουν αλλαγές από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς να ενημερώνονται οι παραγωγοί μας. Χρειάζονται πολλά χρόνια για την προσαρμογή. Γι' αυτό θα ήθελα σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα να στρέψετε την προσοχή σας γιατί είναι μια πολύ σοβαρή απειλή και πραγματική απειλή. Και σίγουρα θα πρέπει και αυτή την πτυχή να τη λάβουμε υπόψη ότι αφορά τη διαμόρφωση του μελλοντικού ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο, ευχαριστώ και όλους όσους πήραν το λόγο και τώρα η υπουργό Έλενα Εσπινόζα έχει το λόγο για να μας πει μερικά πράγματα και τη σκέψη της για την όλη συζήτηση και μετά θα ολοκληρώσουμε και την συνάντηση αυτή. Έχεις το λόγο αγαπητή Έλενα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους σας. Θα ήθελα βέβαια να πω μερικά πράγματα απαντώντας όσα άκουσα εδώ στην ε, ημερίδα εργασία πριν να μπω σε γενικότερες ε, σκέψεις και απόψεις. Κάτι που άκουσα από τον κύριο Μαρτικόλσκι που είπε για το τι ισχύει για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, και μια αναφορά επίσης στην Ισπανία σαν χώρα. Θα ήθελα να σας πω, έστω και αν δεν είμαι εδώ με την ιδιότητά μου σαν Ισπανίδα υπουργό, αλλά σαν προεδρεύουσα των Υπουργών Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, αλλά να σας πω το εξής. Στην Ισπανία ούτε μία περίπτωση διαπιστωμένη δεν υπήρξε καλλιέργειας καλαμποκιού. Και βέβαια σε μέσα ενημέρωση ακούσαμε διάφορες πληροφορίες, αλλά εμείς ε, πάντα αναφερόμαστε στην πραγματικότητα και αυτό είναι το χρέος μας. Επαναλαμβάνω, η πραγματικότητα είναι δεν είδαμε ποτέ καμία διαπιστωμένη περίπτωση παρομοίου προβλήματος. Να σας πω και κάτι άλλο. Τα στοιχεία αυτά βέβαια έχουν ε, προσωρινό χαρακτήρα και όλα τα κράτη-μέλη όταν τελειώσουμε θα μπορούμε να πούμε ότι η Ισπανία είναι η πρώτη παραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε οικολογικά προϊόντα αυτό δείχνει, όπως το είπατε κι εσείς, ότι αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποφελούμε από τη στιγμή αυτή για να υποβάλω και κάποιες προτάσεις. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια εργασία επικεντρώνοντας την προσοχή μας για μια συνύπαρξη σε κοινοτικό επίπεδο και έτσι να δούμε συγκριτικά τι γίνεται κάνοντα σύγκριση ακριβώς ε, των διαφόρων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα, α και στην Ελλάδα Γκαρσία. Λοιπόν, ε, και αυτό προς δύο κατευθύνσεις. Ε, τι μα είπε ότι εδώ και πέντε χρόνια χάσαμε από τα χέρια μας εργαλεία. Ίσως εδώ υπάρχει κάποιο λάθος θα πρέπει να μιλάμε για τουλάχιστον 7 χρόνια. Η τελευταία αλλαγή ήταν η διάμεση μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2003. Και ακόμα είναι σημαντικό αυτό, ευαίσθητο το θέμα του Λευκού Κενού. Και εδώ επιμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι μια κάποια μορφή ανάπτυξης, εξέλιξης ε, αυτού του λευκού διαστήματος ε, και για τα προϊόντα ακριβώ που έχουν ετικέτα τυποποιημένων προϊόντων. Σε... Ξεχωρίζοντας τα από τα ανώνυμα. Και αυτή τη στιγμή τι κάνουμε και στην Ισπανία. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται μετά από την ε, Ευρωπαϊκή με, με, μετά από την κρίση. Είτε καταλαβαίνει κανείς ότι τα ανώνυμα προϊόντα δεν ξέρουμε αν προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις όπως άλλα επώνυμα προϊόντα. Θα πρέπει να δούμε επώνυμα ή ανώνυμα, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή να τα αναλύσουμε εδώ σε ε, αυτό το απόγευμα. Εντάξει, μπορούν να τα δούμε ακριβώς, να δούμε ακριβώς ε, αυτές τα, τις μάρκες, όπως και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Και στην Ισπανία, και με συγχωρείτε που προβάλλω συνεχώς ε, την ισπανική κατάσταση, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, αλλά έχουμε από την ε, Υπουργείο Βημηχανίας Τουρισμού Εμπορίου, έχουμε μια μελέτη και εκεί καταβάλλεται μια προσπάθεια για παράλληλη εξέταση ανάμεσα στην επένδυση που κάνει κάθε βιομηχανικό τομέα στην ε, καινοτομία, ανάπτυξη, έρευνα και τελικά πόσες άδειες εκμετάλλευσης ε, υπάρχουν αναλογικά ή όχι σε σχέση με αυτήν την ε, με αυτά τα χρήματα που δαπανώνται και αν θα πρέπει να δούμε εάν υπάρχει ένα αντίκτυπο ανάμεσα σε αυτά που δαπανώνται και στα, στις καταχωρήσεις μετά, τις προστατευόμενες εδώ. Τη ίδια, ας πούμε, στο, για το ίδιο προϊόν, η ίδια βιομηχανία έχει και το ανώνυμο προϊόν, αλλά έχει και το επώνυμο ε, προϊόν που διαφέρει από το ανώνυμο που θέτει πάλι σε εμπορία. Τι γίνεται εδώ. Χρησιμοποιεί μια διαδικασία και θα μπορούσε να καταγγελθεί αυτό και στα τρόφιμα όπως και στα φαρμακευτικά γιατί υπάρχει κανονικά μια καταχώρηση δήλωση αυτής της επένδυσης. Τι γίνεται, δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Πολλές φορές τα ανώνυμα προϊόντα ε, νομίζω ότι παράγονται από την ίδια βιομηχανία. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε τίποτα περισσότερο. Υπάρχουν ε, πάντω δύο αλυσίδε που παράλληλα εργάζονται ή με το ανώνυμο προϊόν ή με το υπόνυμο. Αυτά ήθελα να πω και να αποφύγουμε κάτι που θα προκαλούσε μια κάποια σύγχυση και θα πρέπει να δούμε περισσότερο γενικού χαρακτήρα δηλώσεις και θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν όλους σας ε, για τα συμπεράσματά σας. Η κτηνοτροφία, η γεωργία, η τεβιμηχανία παραγωγής τροφίμων. Ε, ε, νομίζω υπάρχει ένα πρώην και ένα μετά. Και αυτό έχει σχέση και με τις τρέλες αγελάδες. Και τελικά, τι κάνουμε εδώ συντάσσουμε νέες ρυθμίσεις και να μπορέσει να ισχύσει για κάθε μια δραστηριότητά μας παραγωγής με απαιτήσεις. Μπορούμε να πούμε και μάλιστα υπερήφανα ότι ε, υπάρχει ασφάλεια όσον αφορά αυτή την αθωότητα σε εισαγωγικά και μάλιστα στο 100% των προϊόντων μας και αν για κάποιο τέλο πάντων ελάχιστο λαθάκι βγαίνει ένα πρόβλημα στη μέση που έχει να κάνει και με το σύστημα ανιχνευσιμότητας σε λίγα λεπτά μέσα είμαστε θέση να γνωρίζουμε πού συνέβη αυτό και με ποιο τρόπο πώς. Και αυτό ε, καθησυχάζει και τον ε, καταναλωτή και με συγχωρείτε που δεν θα μιλήσω τώρα σαν ε, προεδρεύουσα, θα μιλήσω σαν καταναλώτρια. Εδώ τι έχουμε συνηθίσει, να μην κινδυνεύουμε από ένα προϊόν. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν το αναγνωρίζουμε αυτό ότι αυτό τι προσπάθεια για να μην διατρέχω κανένα κίνδυνο εγώ σαν καταναλώτρια οφείλεται σε αυτό που έκαναν και οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες και οι μεταποιητές. Και εδώ. Τώρα λέμε τώρα ότι... Ε, εδώ λέμε ότι θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο καταναλωτής. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μιλάμε και για την ε, ευμαρία των ζώων. Και εδώ επιμένω. Εγώ θα είμαι και παρατηρήτρια και πολίτης. Ε, ας πούμε, πάνω χάρη στην ε, τηλεόραση που επηρεάζει περισσότερα τα πράγματα. Όταν βλέπουμε διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, ε, ε, διάφορες, ε, διάφορα κτηνοτροφία, το ένα άλλο, και μας πιάνει μια λύπη για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται κανείς αυτά τα ζώα. Και εδώ έχουμε διαφορετικά που ισχύουν για την αντιμετώπιση, για την τι κάνουμε με τα ζώα και δεν μπορέσαμε δυστυχώς κατά την άποψή μου να το εξηγήσουμε στον καταναλωτή και να του πούμε και αυτό το πληρώνουμε τώρα. Και αν δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι ακόμα πιο δύσκολο ήταν να το κάνουμε πέρα των συνόρων μας των ευρωπαϊκών. Και τώρα Εάν είμαστε απέναντι σε μια αγορά περισσότερο όρημη, τουλάχιστον παρόμοια με την ευρωπαϊκή αγορά, εντάξει αυτό θα ήταν αρκετά εύκολο. Αλλά τι γίνεται σήμερα, μπαίνουμε και σε όριμες ε, αγορές αλλά και σε αναδυόμενες χώρες όπου υπάρχουν διαφορετικές συνήθειες και διατροφής ε, και λοιπά και πολιτιστικές επίσης και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερες δυσκολίες να τα εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα. Υποχρέωση, δεν ξέρω, δεν θα μπορούμε που δεν είναι να γυρίσουμε πίσω για να δούμε πώς θα είναι να πλωστευτούν τα πράγματα, οι ρυθμίσεις για τη μηχανία, για τη γεωργία, για τη διατροφία. Και άλλο όμως είναι πώς ε, θα κερδίσουμε στον τομέα ε, της εξασφάλισης. Ε, τελικά δεν μας συγχωρεί ο καταναλωτής αν πάμε πίσω. Και ας πούμε για τα αυτοκίνητα, τα airbag, η αερόσακη ήταν υποχρεωτική ε, στα αυτοκίνητα και τώρα είναι αδιανόητο να έχουμε αυτοκίνητο χωρίς αεροσακό γιατί ε, όλοι μας ξέρουμε το πώς σιγουριά μας προσφέρει στον δρόμο. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να συνάδουν και με την ανταγωνιστικότητά μας. Και εδώ πιστεύω ότι πολλές φορές διαπράξαμε και εξακολουθούμε να διαπράττουμε κάποια σφάλματα. Σίγουρα, οποιοδήποτε προϊόν εισέρχεται στην Ένωση από τρίτη χώρα, θα πρέπει να υπόκειται σε αντίστοιχες ισοδύναμες απαιτήσει. Είπα, ισοδύναμες απαιτήσεις. Αυτό που είπα στην ομιλία μου είναι ότι χρειαζόμαστε όχι μόνο ισοδύναμες απαιτήσει, αλλά εναρμονισμένες απαιτήσει. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας εξηγήσω αυτούς τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούμε μερικές φορές. Όταν μιλούμε για ισοδυναμία, για αντιστοιχεία. Νομίζω ότι πολύ καλά μας το εξήγησε αυτό, δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Γιάρ, αλλά νομίζω ότι εκείνος το επισήμανε. Όταν μιλούμε για ισοδυναμία, για αντιστοιχεία, εννοούμε ισότητα στο στόχο της τελικής προστασίας. Δηλαδή είναι μια έννοια που είναι προσανατολισμένη προς το στόχο. Αν όμως απαιτούμε εναρμόνιση, μιλούμε για εξ αρχής ταυτότητα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι όμως μόνο προς το τελικό αποτέλεσμα, έχουμε την εναρμόνιση των προτύπων από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα σας το πω με άλλα λόγια που είναι αυτά που χρησιμοποιούμε συνήθως. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να απαιτήσει αμοιβαιότητα σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτει με τρίτες χώρες. Θα ήθελα με αυτό να ολοκληρώσω και να σας ε, πω ότι η εμπειρία μας μας έχει διδάξει ότι έχουμε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο. Ένα μοντέλο που μπορούμε να το υπερασπίσουμε οπουδήποτε στον κόσμο. Έχει μια διαφοροποιημένη ποιότητα αυτό το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Και αυτή η διαφοροποιημένη ποιότητα θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τον καταναλωτή και να πληρώνει και το τίμημα ο καταναλωτής. Σε αυτή την ιδιαιτερότητα οφείλεται η ισχύ μας. Και χάρη σε, αυτή την, αυτό το ενισχυμένο μοντέλο θα μπορέσουμε να ανεφοδιάσουμε γεωργικά προϊόντα όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλες χώρες του κόσμου. Φυσικά όλα θα πρέπει να γίνονται με συνθήκες ισότητας και δυστυχώς αυτή την ισότητα δεν μπορούμε να την απαιτούμε όταν εξάγουμε γιατί εκεί τις, ε, τους κανόνες μας τους επιβάλλουν οι τρίτες χώρες που εισάγουν τα προϊόντα μας. Πάντως, σε ό,τι αφορά την δική μας αγορά, μπορούμε καθημερινά να ενισχύουμε τους κανόνες. Και για το καλό όλων, και εδώ έχουμε μια γενικότερη επισκόπηση, καλύπτοντας ε, το συμφέρον και του γεωργού και του κτηνοτρόφου, μέχρι το συμφέρον του καταναλωτή, όπως είπε η κυρία Γκαρθία Πέρες, θα πρέπει ο γεωργός να ανταμείβεται για το διαφοροποιημένο τρόπο παραγωγής. Αλλά να μην ξεχνούμε και τον τελικό καταναλωτή. Γιατί ο καταναλωτής οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να εγκαταλείψει τα κοινοτικά γεωργικά προϊόντα και να ζητήσει εναλλακτικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να τον κερδίσουν τα δικά μας προϊόντα. Η διαφοροποιημένη ποιότητα είναι πολύ σημαντικό. Η βελτίωση της συχνηλασιμότητας είναι στόχοι που ήδη τους υλοποίησαμε. Τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε την γενίκευση των απαιτήσεών μας για να κερδίσουμε και τις υπόλοιπες αγορές παγκοσμίω και ανεξάρτητα από τις διμερείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που θα πρέπει να περιλαμβάνονται τέτοιες ρήτρε, θα πρέπει να επιβάλλονται τις απαιτήσει. Η νέα κοινή γεωρική πολιτική μετά το 2013 θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο που θα ενισχύει την γεωργία μας. Και η εμπειρία μας σε αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί στην αναγνώριση και τη διόρθωση των σφαλμάτων του παρελθόντος. Γιατί υπήρξαν κάποιες ε, αποτυχίες και λάθη, αλλά από αυτά τα παθήματα θα διδαχθούμε και θα τα μετατρέψουμε σε ισχύ, ώστε η σημερινή απειλή που αντιμετωπίζουμε να μετατραπεί σε ευκαιρία. Πάντως μπορείτε να υπολογίζετε στην Ισπανική Προεδρία, γιατί θα συνεχίσουμε και τώρα να προωθούμε αυτό το θέμα, αλλά και μετά, μετά το τέλος της Προεδρίας μας στο Συμβούλιο Υπουργών. Σας ευχαριστώ θερμά και νομίζω ότι έχουμε μια τεράστια πρόκληση να αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι συναρπαστική για όλους, προκειμένου να εξασφαλίσουμε σε μια όλο και πιο ενωμένη και πιο ισχυρή Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Ελένα Σπινόζα, και την Επίτροπο παρόλο που χρειάστηκε να αποχωρήσει. Α, η κυρία Μαγκίνες θέλει το λόγο. Πρόεδρε, ξέρω ότι είναι αργά. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να κλείσετε τη συνεδρίαση. Αλλά εγώ αναφέρθηκα στι συνομιλίε, την επανεκκίνηση μάλλον των συνομιλιών σε πλαίσιο, στο πλαίσιο τη Μπερκοσούρ. Θα ήθελα μια απάντηση, παρακαλώ. Πρέγω. Σα ευχαριστούμε, κύριε Μαγκίνε. Η Έλενα έχει το λόγο. Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω, να σας δώσω σαν πληροφορία και είναι φρέσκο φρέσκο εδώ και περίπου 24 ώρες ξέρετε ότι πολύ πολύ γρήγορα μπορεί να ξαναλλάξει. Ενδεχόμενα στην επόμενη συνάντηση θα πρέπει να ισχύει η πολιτική συμφωνία για να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή συζητούνται δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα η συμφωνία με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και νομίζω ότι έχει επιταχυνθεί όλη η διαδικασία και επίσης τη συμφωνία Μερκοσούρ όπου η Ισπανική Προεδρία προσπαθεί να πετύχει μια πολιτική συμφωνία έναρξης των ε, διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει εκεί, αλλά ελπίζουμε ναι εμείς. Λοιπόν, αυτά και να έχουν ολοκληρωθεί τα δύο και κάτι λιγότερο μήνες που μας μένουν μέχρι το τέλος τη λήξη της Ισπανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τελειώσαμε και με αυτό. Υκανοποιήσετε και την τελευταία ερώτηση με την απάντησή σας αλλά να τονίσω ότι συμφώνησαν απόλυτα όλοι και έχουν συγκλίνει αυτές οι απόψεις με τις απαντήσεις απόψεις της ε, Υπουργού. Θα σε ευχαριστήσω αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι να μην έχουμε μια στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι παραγωγοί μας να υποφέρουν από ένα παρόμοιο στρεβλωμένο ανταγωνισμό. Επειδή μόνο και μόνο υπάρχουν ορισμένοι που βάζουν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να σέβονται όλα αυτά. Όπως το είπε και η Ελένα αυτό το παράδειγμα του αερόσακου στα αυτοκίνητα δείχνει χαρακτηριστικά την κατάσταση. Δεν θα μπορούσαμε πουδενή να ε, εισάγουμε αυτοκίνητα από τρίτε χώρε χωρί αερόσακο. Το ίδιο λοιπόν γιατί να μην εισηγεί στα τρόφιμα. Εδώ λοιπόν είναι και το θέμα ενημέρωση Θα πρέπει να ενημερώσουμε, να πληροφορήσουμε του καταναλωτέ μα ότι απαιτείται να γνωρίζουν εάν τα προϊόντα αυτά σέβονται τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά, τι περιγραφέ ευρωπαϊκέ Και ακόμα κάτι να πούμε για τη μέθοδο. Καταλαβαίνουμε το ρόλο που παίζουμε εμεί σαν κοινοβούλιο και χάρη στη Λισαβόνα, στη συνθήκη τη θα πρέπει να αντιληφθούμε ακόμα περισσότερο ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνδυασμένα θα μπορούσαν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην νομοθεσία την ευρωπαϊκή. Και όπως απόψε κάναμε εδώ σε αυτή την ομάδα εργασία, προωθώντας, προτείνοντας πράγματα για τον ε, ανταγωνισμό με συγκεκριμένα πράγματα και ο Επίτροπος μας ανακοίνωσε ορισμένες πρωτοβουλίες σημαντικές ε, το φθινόπωρο. Θα πρέπει να δώσουμε ένα ε, καταλάβουν όλοι ότι οι πολίτες τους οποίους εκφράζομαι εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε, να νομοθετήσουμε, να ρυθμίσουμε κατάλληλα. Ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστούμε την Ελά Εσπινόζα της 18 Μαΐου στο Στρασβούργο στις 6, όχι, στις 7 το βράδυ θα συνεχθούμε και πάλι. Γεια σας και ευχαριστούμε. Τελειώσαμε.